Καλό σα απόγευμα κυρίε και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε θα έλεγα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να καλωσορίσω όλου ε, του εξέχοντες συναδέλφου από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μόνοι που παρίστανται και νομίζω ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την θετική παρακολούθηση και συμμετοχή τους και οι άλλες πολιτικές ομάδες ε, προσυπογράφοντας θα ήταν κίνητρο αυτό για αυτές να συμμετέχουν ε, πιο αθρώα στις εργασίες μας. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας, καθώς επίσης και θα συνεχίσει και στη αυριανή συνεδρίαση. Απλά και μόνο για να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω και τους ε, όσους βρίσκονται σε αυτή την κάπως περίεργη αίθουσα εδώ τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής χρειάζομαι και άλλα για να δω που βρίσκονται. Υπάρχει μεγάλος χώρος ε, βέβαια, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταφέρουμε. Τώρα απλά και μόνο για την ημερήσια διάταξη για τις επόμενες δύο ημέρες, αν μπορούμε να εγκρίνουμε αυτή την ημερήσια διάταξη. Η μόνη αλλαγή που έχουμε είναι ότι στις ψηφοφορίες αύριο θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Μπίλαν πριν από του κυρίου Μάιερ την έκθεση αλλαγή στη σειρά. Θα γίνει λοιπόν αυτό αύριο σε σχέση με τις ψηφοφορίες. Στις 10 η ώρα θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε αύριο. Πιο πριν θα έχουμε μια σημαντική παρουσίαση όμως για μια νέα πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση των, όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα που κάπως ε, με καθυστέρηση υποβλήθηκε ώστε να μπορέσουμε λεπτομερώς να την εξετάσουμε σε βάθος. Αλλά από πλευράς ε, των ε, βουλευτών η κυρία Γκέπατ και άλλο συνάδελφο συμμετέχουν ώστε θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θα είναι σημαντικό αυτό. Και ζήτησα από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Εσόδων και από πλευρά ε, αυτή τη διεύθυνση ο κ. Ζελίνσκι θα παραστεί για να δώσει κάποιε επεξηγήσει. Το άλλο θέμα το οποίο πρέπει να ε, ψηφίσουμε προ έγκριση αύριο είναι ένα νέο θέμα. Θα έχουμε ένα διορθωτικό όσον αφορά την ε, πρόταση για τα μέσα και είναι απλά και μόνο μία διόρθωση των ε, προτάσεων του παρατήματος. Αυτό θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη επιπρόσθετα αύριο, τον 10. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επίσης θέλω να υπενθυμίσω Όλα τα έγγραφα αυτής της συνεδρίασης είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όσοι έχετε λοιπόν ηλεκτρονικά μέσα μπορείτε να ε, έχετε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα μέσω των ε, συσκευών σας. Και φυσικά μπορείτε να τα εξετάσετε και όλο και περισσότεροι νομίζω χρησιμοποιούν πλέον αυτά τα μέσα. Δεν θα υπάρξει νέο, ε, νέα επιστολή ενημερωτική, αλλά εκείνη που θα έχουμε για την επόμενη συνεδρίασή μας. Και προτού περάσουμε στα ουσιώδη στοιχεία των εργασιών μας, υπάρχουν πρακτικά που έχουν δημοσιευθεί για την συνεδρίασή μας της 9 η Ιανουαρίου. Και θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται κατά τα τέλη της συνεδρίασης αν δεν έχουν εγερθεί κάποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις από τα μέλη μέχρι τότε. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε τώρα, προτού περάσουμε το θέμα της έκθεσης του καθηγητού Αντώνιο Κορέντε Κάμπος είναι να ζητήσω από τους εισηγητές και άλλους να μας ενημερώσουν για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τους τριμερείς διαλόγους. Με χαρά βλέπω ότι η κυρία Σάντε Μόζα είναι παρούσα εισηγήτρια για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, τον κανονισμό σχετικά. Θα τη ζητήσω σε μια στιγμή να μας ενημερώσει ...στην πρόοδο ή έλλειψη, απουσία πρόοδου, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και ποιες είναι οι προσδοκίες της. Η ε, κυρία Κονελάνεν δεν παρίσταται και μπορώ ίσως έτσι να εξετάσουμε να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες ε, public procurements. Ε, είναι ένα σημαντικό σύντομο κείμενο νομοθετικό Άκρο σημαντικό όμως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε προς την ηλεκτρονική, ηλεκτρονικούς λογαριασμούς. Και η συνάδελφος έχει μεγάλη πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά την, το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και υπάρχουν ε, θέματα τα οποία έχουν ε, γερθεί και εξεταστεί και τώρα έχουμε καταλήξει σε συμφωνία μετά από δύο τριμερείς ε, διαλόγους. Θα θυμόσαστε και το θέμα της εντολής για διαπραγμάτευση. Θα είναι παρούσα αύριο η συνάδελφος για να μας παρουσιάσει αυτή τη συμφωνία. Και έτσι δεν θα εξετάσω αυτά τα σημεία τώρα κατά λεπτέστερα πιο εξειδικευμένα σήμερα το απόγευμα. Απλά και μόνο να πω, α, παρίσταται η συνάδελφος. Θα σταματήσω λοιπόν τώρα εγώ να σχολιάζω και η ίδια μπορεί να μας τα σχολιάσει πιο εξειδικευμένα. Εντάξει λοιπόν. Και από αυτή την πλευρά τώρα είμαστε έτσι. Ωραία. Και μια και, μια και θα ζητήσω από τη συνάδελφο να παρέμβει σε ένα λεπτό, απλά και μόνο να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την πρόοδο για τον δεύτερο τριμερή διάλογο. Για το τελευταίο σημείο του νομοθετικού πλαισίου ως ε, πρόταση για τα για τον εξοπλισμό υπο ε, εργαλείων ε, υποπίεση και δεν ήταν τόσο απλά τα θέματα ε, όσο περιμέναμε. Έκανε κάποιες αλλαγές ε, το Συμβούλιο τα που δεν ήταν ε, αναμενόμενες. Όμως έχουμε μια συμφωνία τώρα σε σχέση με αυτόν τον εξοπλισμό και αυτή η συμφωνία θα τεθεί προς ψήφιση προς έγκριση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με αυτόν τον εξοπλισμό, τα θέματα έχουν προχωρήσει. Η κυρία Κρονλάνγκ, παρακαλώ. Προτού προσέθετε στην αίθουσα, ενημέρωσα ότι θα έπρεπε να υπάρξει πληροφόρηση για το πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχουν προοδεύσει. Εσείς η έχετε τον λόγο να μας τα πείτε παρακαλώ. Συγγνώμη πρόεδρε που καθυστέρησα να προσέλθω. Και δυστυχώς σε σχέση με τα όσα είπατε δεν μπόρεσα να τα παρακολουθήσω, απλά και μόνο πολύ σύντομα. Στον τριμερή διάλογο συμφωνήσαμε η συμφωνία αυτή είναι δεδομένη και διαθέσιμη και όπως προαναγγέθηκε σε σχέση με ε, το πεδίο εφαρμογής οι γενικές απαιτήσει ε, έχουν εξειδικευθεί όσον αφορά τον ε, αμερόληπτο ουδέτερο ρόλο των, της χρήσης των τεχνολογιών και απαρίθμηση των ουσιοδών στοιχείων από πλευράς ηλεκτρονικών εξοπλισμών, σε, από πλευράς άρθρων ε, μέσα σε μια περίοδο 36 μηνών θα πρέπει η περίοδος δοκιμασίας ε, να έχει ολοκληρωθεί και να έχει προχωρήσει όσον αφορά την ε, δυνατότητα ε, αξιοπιστίας και λειτουργικότητας αυτών των εξοπλισμών. Ε, η δυσκολία ήταν η περίοδος εφαρμογής 18 μήνες όσον αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες και 6 μήνες παραπάνω για τις υποδέστερες ε, αρχές. Ε, νομίζω αυτό είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο που κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες όσον αφορά τον χρονορίζοντα για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και κατάφερε να πείσει το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ξέρετε, εγώ ακολουθώ εντολές. Νομίζω ότι πολύ καλά τα καταφέραμε και εσείς και οι σκιώδεις εισηγητές. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο. Και τώρα, για να ολοκληρώσουμε με αυτή την ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους, θα παρακαλέσω την κυρία Σάλντε Μόζη για να μας πει και αυτή που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των καταναλωτικών πρώτων και φαντάζομαι θα μιλήσετε για την εποπτεία των αγορών. Σάλντε Μόζε, ναι, πράγματι θα καλύψω όλη αυτή τη δέσμη. Στη Δανία λέμε no news, good news. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε καμία είδηση από το Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν είναι καλή είδηση. Θεωρούμε ότι είναι κακή είδηση στην προκειμένη περίπτωση. Θα ήθελα να είμαι πολύ ξεκάθαρη. Δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο πριν τα τέλη δυστυχώ αυτή τη κοινοβουλευτική περίοδου. Έπαψαν το, πιστεύω, ότι μπορούσαμε να το πετύχουμε. Τώρα λοιπόν αυτό το οποίο σχεδιάζουμε είναι να κατεβάσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια και συζητάμε το χρονοδιάγραμμα. Ποιο θα ήταν ε, το καλύτερο timing. Διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε αρκετό χρόνο και για να διεξαγάγουμε μια καλή συζήτηση και βέβαια και μετά θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ε, μια στο δυνατόν ε, πιο μια ολομέλεια πιο αργά. Ο Απρίλιος όμως είναι πολύ φορτωμένος. Τέλος πάντων το επεξεργαζόμαστε ακόμη το θέμα, δεν έχουμε επιλέξει την ολομέλεια στην οποία θα προσπαθήσουμε να συζητηθεί το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε όμως την κατάλληλη χρονική στιγμή. Όταν θα γνωρίζω περισσότερα θα σας ενημερώσω. Και φυσικά όταν γνωρίζω οτιδήποτε και για την ημερομηνία... Εγώ το ο σπιτικά είναι εννοώ βέβαια, έτσι. Θα σας ε, ενημερώσουμε, θα ενημερώσουμε καταρχάς τους κοιόδες για να συζητήσουμε μαζί το πώς θα προχωρήσουμε και ίσως ε, να καταλήξουμε σε νέους συμβιβασμούς. να δούμε αν θα αλλάξει έκθεση ή όχι. Ακόμη είναι ανοιχτό το θέμα. Αλλά όταν θα είναι γνωστή η ημερομηνία τη ε, συζήτηση στην Ολομέλεια και τη ψηφοφορία, τότε θα τα συζητήσουμε αυτά. Αυτά λοιπόν ε, είναι τα νέα μα, δηλαδή καθόλου νέα επί τη ουσία. Πρόεδρο. Πράγματι το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετέ φορέ. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε την απογοήτευση του ότι δεν καταφέραμε να έχουμε κάποια εξέλιξη. Λάβουμε υπόψη μας ότι ψηφίσαμε τον Οκτώβριο την έκθεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ολομέλεια, είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τις πολιτικές ομάδες ε, για να δούμε την ημερήσια διάταξη. Κατά την άποψή μου, αν θέλουμε να βρούμε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για να συζητηθεί και να συζητηθούν μάλιστα και οι δύο προτάσεις, η πιο ρεαλιστική ημερομηνία είναι ή η Ολομέλεια του Μαρτίου στο Στρασβούργο ή η μήνυ Ολομέλεια στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο. Επειδή μαζεύονται πολλά στο τέλος, μιλήσαμε και με τη διάσκεψη των πρώτων των επιτροπών στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και ενημερώσαμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Μπορεί να χρειαστεί να, περικοπούν, να περικοπεί ο χρόνος συζήτηση επειδή θα είναι πολλές οι προτάσεις που θα συνοστιστούν στο τέλος θα δούμε τι θα αποφασίσουν και οι γραμματείες των πολιτικών ομάδων. Πρέπει να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ και θα περάσουμε τώρα στην εξέταση ε, του σχεδίου έκθεσης ε, για την ε, πρόταση κανονισμού για την αμοιβαία συνδρομή των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και συνεργασία αυτών με την Επιτροπή. Αντώνιο Κορέντε Κάμπο είναι εισηγητή μα. Να καλωσορίσω και τον κύριο Ρο. Πρόσφατα ήλθε εδώ. Χαίρομαι διότι έδειξε σύνεση και σας έδωσε το ελκθέσει εδώ. Βλέπω και τον Όλε Σμίτ από του Φιλελευθέρου. Ε, βλέπω την Άσλι Φόξ, μάλλον τον Άσλι Φόξ. Α, η κυρία Μακλάρκ θα είναι στη θέση του. Από του πρασίνου δεν υπάρχει κανείς προς το παρόν, αλλά ας ακούσουμε καταρχάς τι έχει να μας πει ο εισηγητή ή σκιώδη εισηγητή, τες και όποιο άλλος συνάδελφο θέλει το λόγο. Τώρα ψάχνω και την Επιτροπή. Μάλιστα, εκεί πίσω είστε, οκ. Okay. καλά σας... Ε, Ξενάκης, δυστυχώς δεν μπορεί, <laughs> δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Διορθώνει μου λέει τη σωστή προφορά ο συνάδελφος δίπλα που είναι Έλληνας. Λοιπόν, θα σας δώσουμε το λόγο μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Okay. Ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, η δράση κατά της παραβίασης ε, της τελωνικής νομοθεσίας έχει θεμελιώδη σπουδαιότητα για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αλλά όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και την ανάπτυξη της τελωνιακής συνεργασίας. Υπάρχει ένας κανονισμός ε, του 1997, αλλά που υπάρχουν κενά και δημιουργούν ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά και ανησυχητικών διαστάσεων, σύμφωνα με τη μελέτη επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση. Οι τελωνιακοί φορείς δεν έχουν μέσα για να ανακαλύπτεται αν τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται ανταποκρίνονται στην πορεία την διαδρομή ενός εμπορευματοκιβωτίου και σε σχέση με το καθεστώς μετακομιστικού εμπορίου, σε σχέση και με τις διαδικασίες αυτές. Το 2011 τα κράτη-μέλη ανακοίνωσαν ε, χίλιες τόσες περιπτώσεις όσον αφορά παρατυπίες και για ένα ποσό 108 εκατομμυρίων ευρώ απολειών που συσχετίζονται με την ε, παραπλανητική περιγραφή των εμπορευμάτων. Πρόκειται για απώλειες που αφορούν τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Το, οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος όμως είναι μεγαλύτερες. Οι περιπτώσεις παραβίασης όσον αφορά το διαμετακομιστικό εμπόριο πλησιάζουν τις ε, απώλειες ε, ε, εκατομμυρίων ευρώ ανά έτοσα και δεν υπάρχουν στοιχεία επαρκή για χιλιάδες περιπτώσεις ενδυνάμει απατών. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις, όσον αφορά τις εξεταστικές ενέργειες της ΟΛΑΦ, η περίοδος ε, μέχρι 7 μήνες όσον αφορά τον έλεγχο των εγγράφων εισαγωγών, εξαγωγών, είναι μια σημαντική πηγή απολειών. Το ελεγκτικό συνέδριο το 2010 σε ελεγκτικές ε, ε, δράσεις είπε ότι σε μια δειγματοληπτική δράση βρέθηκαν 49 σφάλματα τα οποία εκπροσωπούν άμεση απώλεια του ύψους ε, πάνω από μισό εκατομμύριο, πάνω από 500.000 ε, ευρώ. Αυτά τα ποσά μπορεί να παραγραφούν και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να ανακτηθούν σε σχέση με τον προϋπολισμό της Ένωσης. Δεν εισπράττονται λοιπόν μια και η παραγραφή μπορεί να ε, δώσει συνέχεια στην περίπτωση αυτή των απατών και σε σχέση με την έκθεση που σας υποβάλλω, ε, το θέμα είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε ώστε να καταπολεμηθούν αυτές οι απάτες, ε, τελωνιακές απάτες και να ε, ενδυναμωθεί η ασφάλεια στην εσωτερική αγορά σε σχέση με τα προϊόντα που διακινούνται και να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Διότι η αύξηση των απατών απαιτεί μηχανισμούς πρόληψης και καταπολέμησης και στο επίπεδο των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου εδώ μια σύντομη παρατήρηση για τις ε, ουσιώδεις, ε, ουσιοδέστερες τροπολογίες που κατέθεσα. Η 6 για ε, να μπορεί να συνάδει με τους ορισμούς στο πρώτο άρθρο για να υπάρχει αντιστοιχεία με τα υπόλοιπα στον κανονισμό γίνεται μια επεξήγηση σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τον ιδιωτικό και τον δημόσιο Υπάρχει εδώ και η αναγνώριση όσον αφορά τις διαδικασίες για την νομική και ε, νομοθετική ασφάλεια σε σχέση με τις, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να μπορούν να γίνονται αποδεκτά από τα κράτη-μέλη αμοιβαία και προτείνεται να παρατείνεται η δυνατότητα της αρρωγής αυτής ώστε να μπορεί να διαφοροποιείται το καθεστώς αυτό. Στο, άρθρο, στο αντίστοιχο άρθρο για τη συλλογή των στοιχείων αν έχουμε μόνο τα εμπορευματοκιβώτια τα οποία διακινούνται ε, στο διαμετακομιστικό εμπόριο μέσω των πλοίων θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής ε, όσον αφορά και την ε, μεταφορά είτε εναέρια είτε και χερσαία στο ε, επόμενο άρθρο για τα διατακτικά δεν συμπεριλαμβάνεται ένα καθεστώς προστασίας ε, δεδομένων γιατί δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα τα οποία να συμπεριλαμβάνονται. Δεδομένων λοιπόν των ανησυχιών που κατατίθενται σε σχέση με την προπαρασκευή αυτής της νομοθετικής πρότασης θεωρούμε ότι πρέπει ρητά να διευκρινιστεί ότι δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται εδώ οποιοδήποτε στοιχείο προσωπικού χαρακτήρα. Τροπολογής 22-23 για το αντίστοιχο άρθρο όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του νέου άρθρου θα πρέπει να τονιστεί η ευθύνη των κρατών μελών να παρέχουν τα στοιχεία αυτά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ζητούνται αυτά από την Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη ή οι οικονομικοί φορείς είναι αρμόδια να παρέχουν αυτά τα στοιχεία όπως ζητούνται και απαιτούνται. Και δύο εβδομάδες μετά από το αίτημα όταν αυτό διατυπώνεται, τι συμβαίνει. Τα κράτη-μέλη δεν απαντούν τώρα, δεν δίνουν τις ε, σε σχέση με τα αιτήματα αυτά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πράγμα το οποίο δεν δίνει δυνατότητα να συνεχιστούν οι ε, εξακριβώσεις. Γι' αυτό θα πρέπει μέσω της δράσης των κρατών μελών και μετά από περίοδο δύο εβδομάδων να έχει τη δυνατότητα άμεσα να ε, ζητήσει από αυτούς τους παρόχους αυτά τα στοιχεία ώστε να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος τέτοιων περιπτώσεων απατών η περίοδος δύο εβδομάδων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να ε, διευθετούνται αυτά και αν δεν υπάρξουν ε, απαντήσεις ε, τότε σε σχέση με ένα άμεσο αίτημα ακριβώς σε σχέση με ένα άμεσο αίτημα αυτεπάγγετα δηλαδή θα μπορεί να υπάρχει δράση. Εδώ έχουμε μια σημαντική σημείωση. Εφιστούμε την προσοχή σε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη μετάφραση στα αγγλικά και στα ολλανδικά τουλάχιστον από τα όσα μπόρεσαν να εξεταστούν σε σχέση με τις μεταφράσεις. Υπήρξε μια κακομετάφραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δίνει συνέχεια στα αιτήματα όλων των κρατών μελών και όχι μετά από αίτημα από κράτη-μέλη όπως βρίσκεται στο κείμενο το οποίο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Εδώ σε σχέση με αυτή την ε, φράση θα πρέπει να, ε, το ένα α να ισχύει σε σχέση με το δεύτερο εδάφιο. Και εδώ υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα 1α και όχι 10. Και σε σχέση με την τροπολογία για την διόρθωση έχει προβλεφθεί αυτό. Για την επόμενη περίπτωση από πλευρά τροπολογία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να έχει την δυνατότητα να δέχεται έγγραφα από τρίτε χώρε στα οποία πρέπει να αναγνωρίζεται, να δίνεται το ε, επίπεδο εκείνο το, να αναγνωρίζεται και δεν ε, χρειάζεται να ζητείτε μία ε, μετάβαση ε, σε άλλη έδρα, πράγμα το οποίο απαιτεί πρόσθετα έγγραφα. Μια και αυτά τα έγγραφα μπορούν με ένα πιο απλό τρόπο, πιο οικονομικό τρόπο να διαβιβάζονται και να γνωστοποιούνται. Οι τροπολογίες 29 και 30 στο άρθρο 31 για τις προθεσμίες και τις, ε, τα στοιχεία αυτά και για την απάντηση από πλευρά των κρατών μελών ή των οικονομικών φορέων. Όταν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε σχέση με τις ε, ε, σύντομες προθεσμίες τριών και πέντε ετών που προβλέπονται ε, από τον ενισχύ κανονισμό. Από αυτή την περίοδο θα πρέπει μέχρι 7 χρόνια να παρατείνεται η περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων ώστε να αποφεύγουμε τον κίνδυνο της παραγραφής. Εδώ υπάρχει ένα σύνολο λοιπόν τροπολογιών όσον αφορά την προστασία δεδομένων και θεωρούμε ότι πρέπει να απλουστευτεί το κείμενο αν είναι δυνατόν. Αυτή η απλούστευση θα μπορεί να δίνει και μια καλύτερη ερμηνεία του κανονισμού χωρίς να υπάρχουν περιττές επαναλήψεις ε, και να υπάρχει διαρκής αναφορά και επανάληψη σε σχέση με τα στοιχεία του κανονισμού υποχρεωτικής εφαρμογής. Και θα ήταν λοιπόν ε, ε, πραγματικά περιττό να επαναλαμβάνονται τέτοιες διατυπώσεις όπου δεν χρειάζονται. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι μετά από δύο μέρες, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου. Η συζήτηση, η εξέταση και η ψήφιση θα γίνει τον Μάρτιο. Και αν όλα πάνε σύμφωνα με τα όσα προβλέπουμε θα περάσουμε στην Ολομέλεια περίοδο συνόδου του Απριλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ σαφή αυτή παρουσίαση. Είναι πάντοτε δύσκολο να ασχολείται ένας εισηγητής με τροποποίηση και τροπολογίες ενός κανονισμού γιατί πρέπει να κατανοήσει και τον νομικό κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και δίνω τώρα το λόγο για σχόλια στους σκιώδεις. Ο κύριος Ρος καταρχάς. Ε, Mr. President, uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των επιχειρήσεών μας και βέβαια και τα συμφέροντα και των καταναλωτών μας θα πρέπει να υπάρχει απλούστευση του κανονισμού για τα τελωνία και συνεργασία μεταξύ των εθνικών τελωνιακών αρχών. Γι' αυτό και θα πρέπει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα για να αποτρέπουν τις παραβάσεις των ελληνικών διατάξεων. Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή, ωστόσο εδώ ε, θέλω να κάνω κάποια σχόλια, να σας περιγράψω τις πιο σημαντικές μου σκέψεις. Σε ό,τι αφορά αυτό το ευρετήριο στοιχείων, η τροπολογία 8 και η τροπολογία 16 είναι σημαντικές. Πρέπει να είναι ε, αυτές οι απόρριτες πληροφορίες να προστατεύονται. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες και για τα σφαίρα των κρατών μελών. Υπάρχει τροπολογία 19, 20, 21 όπου ο εισηγητής ε, τροποποιεί άρθρα τα οποία άπτονται της προστασίας των δεδομένων. Συμφωνώ ε, επί της ουσίας, γιατί είναι τεχνικές πιο πολύ αλλαγέ, αλλά αυτό που θέλω να εξασφαλίσουμε είναι να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον ε, προβλήματα με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Διότι αυτό φοβάμαι. Τροπολογία 22 και 23 σε ό,τι αφορά την δυνατότητα η Επιτροπή να λαμβάνει από τους οικονομικούς παράγοντες απευθείας πληροφορίες. Το θέμα είναι λεπτό. Διότι αφενός θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, αλλά αφετέρου έχουμε και τις επιχειρήσεις μας. Πώς θα σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας αν αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει ε, στις επιχειρήσεις μας. Ενδιαφέρουσα μένει η προσέγγιση του εισηγητή, όμως οι καταναλωτές θα προστατεύονται, αυτό είναι το ερώτημα. Και ολοκληρώνω με την περίοδο αποθήκευσης ε, των ε, δεδομένων και την βάση ΦΙΝΤΕ. E. Έχουμε εδώ επιμήκυνση της προθεσμίας. Μιλάμε για διοικητικές έρευνες, ποινικέ ε, έρευνες. Η προτινόμενη επιμήκυνση δεν μου φαίνεται απαραίτητη. Τρία και έξι χρόνια είναι τώρα η προθεσμία. Νομίζω ότι είναι αρκετή. με τον κύριο Ντεκάμπος και άλλους συναδέλφους βέβαια έχουμε συζητήσει ε, το θέμα και θα το συζητήσουμε και τις επόμενες εβδομάδες και δύο αυτές τις προτάσεις που σας έκανα. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε ρό. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά κύριε Κορέα. Και είπε και ο πρόεδρο ότι υπό τι παρούσε συνθήκε ε, δεν ήταν εύκολο το έργο σας. Φυσικά έπρεπε να δράσουμε γρήγορα, διότι αλλιώ δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι επίκαιρο και είναι και άκρο πολιτικό το έγγραφο. Αφορά πόρους οικονομικούς, αφορά, αφορά την απάτη, αφορά και τη διαφθορά θα έλεγα εγώ. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε διαβάσει την έκθεση ε, της προηγούμενης εβδομάδας, όπου η Επίτροπος Μάλστρομ δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μέσος όρος ε, των πολιτών ε, και μάλιστα που πιστεύουν δηλαδή ότι υπάρχει διαφθορά είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι 6%. Δεν ξέρω. Για τη Βρετανία ίσως θα ήταν ε, πιθανό, αλλά με εξέπληξε, με εξέπληξε που είδα και για τη χώρα μου τόσο υψηλά ποσοστά. Να πιστεύει ο πολίτη δηλαδή ότι υπάρχει διαφθορά και απάτη. Έτσι έχουν τα πράγματα όμως. Και γι' αυτό, πώ να το πω, πρέπει να δράσουμε κατά τρόπο ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πάντοτε πίστευα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι άλλο είναι αν δεν είναι τελωνιακή ένωση, αφού από αυτό ξεκίνησαν όλα. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, και αγαπητή, ο αγαπητός συνάδελφος το έθεσε το θέμα της επικουρικότητας, Είναι σαν μια κίτρινη κάρτα που την δείχνουμε έτσι πάρα πολύ εύκολα. όταν είναι μια λέξη που ακούγεται συχνά, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση τη αρχή επικουρικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Η Κομισιόν και ο Όλαφ πρέπει να έχουν στη διάθεσή του ε, ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση τη απάτη και θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίε άμεσα από του οικονομικού φορεί. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το εδάφιο του κειμένου. Πράγματι είναι λεπτό το θέμα, συμφωνώ. Όμως κάτι πρέπει να κάνουμε. Χάνονται πάρα πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Η πρόταση του εισηγητή είναι να ενημερώνονται δύο εβδομάδες ε, νωρίτερα τα κράτη-μέλη. Ναι, δεν είναι και κακό. Καλή συμφωνία είναι αυτή. Ιδίω αφού τα θέματα που ρυθμίζονται με την έκθεση αυτή είναι και τα θέματα της συνεργασίας ε, μεταξύ κρατών μελών και κομισιών, όχι μεταξύ οικονομικών φορέων και κομισιών. Όπως είπα όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι τους ε, αφήνουμε χαλαρούς πολλές φορές. Οπότε σκέφτομαι να καταθέσω κάποιε τροπολογίες από αυτού. Βέβαια πάντοτε θα πρέπει να τύχουν και τις σύμφωνες γνώμες των υπολείπων. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή σε ό,τι αναφορά τη μνήα της οδηγίας ε, για την προστασία των δεδομένων και ο κύριος Ρώστο ανέφερε. Ίσως ε, να μην είναι απαραίτητο, ωστόσο θα πρέπει να έχουμε κανόνε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. το θέμα δεν είναι τόσο αν θα έχουμε προβλήματα μετά με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά το αν θα έχουμε προβλήματα με τους πολίτες μετά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους διακανονισμούς και τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή δεδομένων, δεν νομίζω ότι είναι επαρκή τα όσα ισχύουν. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων και με ποιου οργανισμούς, με ποιε οργανώσει. Αυτά θα πρέπει να ορίζονται με πολύ σαφή τρόπο, γι' αυτό και υποβάλλω σχετικέ τροπολογίε. Κατά τα λοιπά, Κύριε Ντεκάμπος, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και ελπίζω να στεφτεί με επιτυχία για να κλείσουμε το θέμα αυτό τον Απρίλιο. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συμβολή σας. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή. Ίσως ε, θα χρειαστεί να μην να είμαστε φονταμεταλιστές ή μη φονταμεταλιστές, αλλά να ακολουθήσουμε μια πιο νεοφιλελεύθερη προσέγγιση στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, ε, κυρία Μακλάρκη νομίζω έχει μπροστά της ε, την παρέμβαση του κυρίου Φόξ. Και αν δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, μετά θα λάβει το λόγο η Κομισιόν. Κυρία Μακλάρκη, όμως. Ναι, μου ζήτησε να πω ο κύριο Φόξ ότι συμφωνεί με το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης ε, του εισηγητού και τον ευχαριστεί που τονίζει ε, την έκταση της τελωνιακής απάτης και τις οικονομικές απώλειες και σε ό,τι αφορά τη διαμετακόμιση και τα σχετικά δεδομένα. Πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, επίσης πολύ πιο προσεκτικά και θα πρέπει στο, στο όσο πιο πρώιμο στάδιο να μπορεί η Κομισιόν να παίρνει σχετικέ πληροφορίες. και μόνο κατόπιν ετοίμως από τα κράτη-μέλη να παίρνουν ε, τα στοιχεία αυτά οι Κομισιόν από τους οικονομικούς φορείς. Δεν συμφωνεί ο κύριος Φόξ ότι θα θεωρείται σιωπηρή έγκριση το αν δεν συμμορφώνεται κάποιος με αυτό το αίτημα. Ο τίτλος της έκθεσης, σύμφωνα με τον κύριο Φόξ, αναφέρεται ρητά στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και κομισιών. Και δεν θα πρέπει η Κομισιόν να προσπαθήσει να υπονομεύσει τη συνεργασία τη με τα κράτη-μέλη, χωρί ρητή δηλαδή έγκριση από τα κράτη-μέλη και να έρχεται σε απευθεία επαφή με του οικονομικού φορεί. Πρέπει επίση να υπάρχουν ασφαλιστικέ ε, δικλείδε για να ρυθμίζεται η πρόσβαση και η διόρθωση στοιχείων που έχουν δώσει τα ίδια τα άτομα ε, που τους αφορούν αυτά τα στοιχεία και θα πρέπει να μην είναι πιο δαπανηρή η διαδικασία από αυτή που προτείνεται. Φυσικά και θα συνεργαστεί με τους ε, σκιώδες εισηγητές για μεγαλύτερη διαφάνεια, ο κύριος Φόξ δηλαδή, και λιγότερη απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ε, τις πολιτικές ομάδες. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Αν όχι, θα δώσουμε πολύ μεγάλη χαρά το λόγο καλωσορίζοντας τον πρόσωπο της Κομισιόν από την Όλαφ. Νομίζω είστε για πρώτη φορά εδώ στην Επιτροπή μας. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο για να σχολιάσετε την ε, πρόταση και τις προτάσεις του εισηγητή. Thank you. <coughs> Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και όντως είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι ενώπιόν σας και είναι ιδιαίτερα μεγάλη η ικανοποίησή μου για το λόγο αυτό και ευχαρίστως ε, θα σχολιάσω την, ε, το σχέδιο εκθέσεως του ε, εισηγητού που υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν στα ουσιώδη της σημεία. Επίσης ε, το άλλο που δίναμε να πω είναι ότι για την πρόταση αυτή που είναι σημαντική για τον αγώνα κατά των απατών στον τελωνιακό χώρο, το σχέδιο εκθέσεως του εισηγητού ενισχύει την προστασία κατά της απάτης καθώς και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων της Κομισιόν. Δεν θα επισέλθω ξεχωριστά στις διάφορες προτάσεις του, θα έρθω σε λίγες από αυτές σε ό,τι αφορά την συνεκτικότητα της ε, προτάσεως για το 18 σε το δικό μας για δεδομένα στην βάση δεδομένων για πληροφορίες εμπορευματοκιβωτίων. Αυτό είναι σημαντική πληροφορία, ενισχύει την συνεκτικότητα και αποκαθιστά ένα σύνδεσμο μεταξύ της μελλοντική ε, βάσης δεδομένων και της υφιστάμενης. Άλλο σημαντικό είναι ότι ο εισηγητής σημείωσε έναν αριθμό διατάξεων που έλειπαν από την πρόταση, όπως για παράδειγμα το 16α το οποίο ενισχύει την ε, διάταξη για το παραδεκτό των αποδείξεων που έχουν αποκτηθεί με δικαστική συνδρομή, με αμοιβαία συνδρομή, τέλο πάντων. Σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί ότι το σχέδιο προτάσεως είναι στραμμένο προς το μέλλον. Βάζει την βάση δηλαδή για την συμπερίληψη των αναλύσεων και πέρα από τις θαλάσσιες μεταφορές για να επεκταθεί δηλαδή η ισχύς προτάσεως και στις ενέργειες και στις θαλάσσιες μεταφορές, και στις χερσαίες μεταφορές, συγγνώμη. Ανοίγει δρόμους λοιπόν για το μέλλον. Και με την έννοια αυτή πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο. Επίσης επιφέρει μια διευκρίνηση ο εισηγητής στο 18 age το δικό μας άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που διατηρούν οι οικονομικοί φορείς. Κατανοώ βεβαίω την συζήτηση και ενδεχομένως τις ενστάσεις των χωρών μελών για αυτή την άμεση πρόσβαση. Βέβαια δεν τους αρέσει να ξεπερνούμε, να ε, υπερβαίνουμε τις αρμοδιότητές τους. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η πρόταση του εισηγητού αποτελεί εύλογο συμβιβασμό μεταξύ των όσων είναι αναγκαία και εκείνων των στοιχείων που ενδέχεται οι χώρες μέλη να αποδεχτούν. Καλό συμβασμό δηλαδή, διότι σημαίνει ότι οι χώρες μέλη θα εμπλέκονται και αυτές στην διαδικασία αυτή αναζήτησης δεδομένων από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς για δεδομένα που χρειάζονται να γνωρίζουν. Ας με επιτρέψετε να απαντήσω στο σχόλιο του κ. Ρος. Δεν νομίζω, η Κομισιόν δηλαδή δεν θεωρεί ότι τίθεται θέμα επικουρικότητας εδώ για τον απλό λόγο. Ως εξή, η δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα ή σε άλλα δεδομένα των οικονομικών ε, φορέων υπάρχει ήδη στη βάση κανονισμού του 1996, του 21-25-1996, που επιτρέπει στην Κομισιόν να εκτελεί επιτόπου ελέγχους και επιθεωρήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι η Κομισιόν έχει ήδη την δυνατότητα να αποκτήσει τα έγγραφα ευθέως από τους οικονομικούς φορεί, βέβαια με τη συνεργασία των χωρών μελών. Δεν είναι όμως απόλυτα υποχρεωτικό να λάβει την έγκριση των χωρών μελών. Η ιδέα είναι να, αντί να στέλνουμε τώρα δύο ανθρώπους, για παράδειγμα στην Ιταλία, στην Ιταλία, στη Φιλανδία, για να πάρουν τα έγγραφα και να πληρώνουμε 5.000 ευρώ και πολλές ανθρωποημέρες, είναι πολύ πιο λογικό να μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή και να λέμε χρειαζόμαστε το τάδε έγγραφο, δώστε το μας. Δεν είναι θέμα επικουρικότητας, διότι το δικαίωμα είναι ήδη και εκτιμένο. Δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου χωρίς να αναφέρω τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλει ο εισηγητής για την απλούστευση του κειμένου. Γνωρίζουμε όλοι πώς συντάσσονται τα έγγραφα αυτά εντός των πλαισίων των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον βαθμό περιπλοκότητας που προκύπτει από τις διαβουλεύσεις και από την επιθυμία των ενδιαφερομένων μερών να είναι τα κείμενα απολύτως ακριβή. Ωστόσο ο εισηγητής κατάφερε να εντοπίσει έναν σημαντικό αριθμό επαναλήψεων με την έννοια ότι υπάρχουν τμήματα του κειμένου τα οποία επαναλαμβάνουν υποχρεώσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν μέσα στον κανονισμό προστασίας των δεδομένων. Ο κανονισμός υπαριθμών 45, ο οποίος ούτως ή άλλως εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να επαναλαμβάνονται παραθέσεις από το κείμενό του σε τούτο εδώ το νομοθέτημα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για τις προτάσεις απλουστεύσεως του εισηγητού σας. Και θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την βαθιά κατανόηση των λεπτομεριών των θεμάτων, διότι είναι πραγματικά τεχνικά θέματα και συχνά, ακόμα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε το πρόβλημα της μη κατανόησης από άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί χρειάζεται βέβαια να του εξηγήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ ιδιαίτερα την ικανότητα που επέδειξε ο εισηγητή σα για να κατανοήσει το κείμενο και να κάνει τι σχετικέ τροποποιητικέ προτάσει οι οποίες ενισχύουν την προστασία της ενιαία αγοράς και των οικονομικών συμφερόντων της ε, ενώσεως απέναντι σε απάτες στα ε, τελωνία ή γύρω από τον τελωνιακό χώρο. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα πάλι στον εισηγητή για να μπορέσει να συνοψίσει τη συζήτηση και να προσθέσει ενδεχομένως σχόλια. Το δε χρονοδιάγραμμα ως έχει ισχύει. Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σκιώδεις εισηγητές που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφεραν να διεισδύσουν στην ουσία, στον πυρήνα αυτού του πολύ περίπλοκου ε, ζητήματος ε, αλλά που έχει τεράστια σπουδαιότητα για την ε, προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών μας. Πολλές φορές παραπονούμαστε πολύ και όταν επισκεπτόμαστε άλλες χώρες, ε, Πρόεδρε, και συμμετείχα και σε μια τέτοια αποστολή και παρακολουθούμε και ακούμε παράπονα συναδέφων, βουλευτών για ατελωνιακές απάτες και για τη διαφορά μεταξύ του δεδηλωμένου περιεχομένου και του πραγματικού περιεχομένου. Πρέπει να καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε την, τα παράπονα αυτά και να περάσουμε στη δράση και σε συγκεκριμένες πράξεις. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι οι τελωνιακές απάτες αποβαίνουν εις βάρος των χρηματοδοτήσεων της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε διαρκώς να λέμε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να βρεθούν μηχανισμοί χρηματοδότησης, πρόσθετης χρηματοδότησης και αηφόρου βιώσιμης ε, ε, χρηματοδότησης και μετά όταν έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό στα χέρια μας να μην κάνουμε τίποτα, να μην κάνουμε τα πάντα για να βελτιω... βελτιστοποιείται αυτός ο μηχανισμός. Και αυτή η στόχη είναι σημαντική. Πρώτον, προάσπιση και υπεράσπιση των καταναλωτών. Να ξέρουμε ότι τα εμπορευματοκιβώτια περιέχουν αυτό που περιγράφεται στα έγγραφα. Και δεύτερο στόχο, ο στόχο να υπάρχει χρηματοδότηση, να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ένωση. Οι συνάδελφοι, ο συνάδελφο Ρο ε, που ανέφερε ε, και είναι χρήσιμα τα στοιχεία αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και μας δίνουν τη δυνατότητα να εξετάσουμε πιο εξειδικευμένα αυτά τα θέματα και θέματα ε, προσωπικής φύσης. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που που είχαμε στις ε, επιτροπές Άγκρη και Λίβε σε σχέση με την ε, οποιαδήποτε σύνταξη έκθεσης γνωμοδότησης ε, δεν θεώρησαν αναγκαίο να γίνει κάποια τέτοια γνωμοδότηση. Και η σημαντικότερη διαφωνία του συναδέφου Ρος αφορά την άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες του παρόχου, του φορέα και εδώ δεν είναι το θέμα της υπαναχώρησης ε, ή ανταπόκρισης. Το θέμα είναι η συνδιαλλαγή με το κράτος μέλος. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε οι απαντήσεις ε, να καθυστερούν και να συνεχίζουν να καθυστερούν επί μήνες όταν μπορούν ε, σε συντομότερες προθεσμίες να είναι διαθέσιμες, να είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία. Συσσωρεύονται όλα αυτά. Οι μήνες για να απαντήσουν γίνονται χρόνια και μετά υπάρχει η δυνατότητα παραγραφής ε, έναντι των ε, όσων έχουν ε, διαπράξει αυτά τα δικήματα. Και συνεχίζονται οι παραβιάσεις. Λοιπόν, ε, ολοκληρώνω λέγοντας ότι στα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, γι' αυτό προτείνουμε μια συμβαστική τροπολογία. Αλλά είμαστε απόλυτα ανοιχτοί από πλευράς ε, αντιμετώπισης να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις προτάσεις ε, των συναδέφων και οδών εισηγητών για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον κυριότερο στόχο. Για τα τρία ή έξι χρόνια, αντί τα πέντε ή και εφτά, ομολογώ ότι είναι ένα θέμα τεχνικού χαρακτήρα αυτό περισσότερο και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία χωρίς δυσκολίες και επ' αυτού. Ο συνάδελφος Σμιτ, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τις προτάσεις του συνάδελφου Σμιτ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χωρίς ε, ακραίες θέσεις και φονταμενταλιστικές θέσεις πρέπει να μπορούμε να εργαστούμε. Και για τις προθεσμίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για από πλευράς Όλαφ, πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε στοιχεία τέτοια στη διάθεσή μας, το δυνατόν αμεσότερα από τους ε, φορείς. Δύο εβδομάδες είναι ένας ε, νομίζω ισόρροπος, ισορροπημένο συμβιβασμός. Αλλά μπορούμε να το δούμε αυτό. Η προστασία δεδομένων. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η προστασία δεδομένων δεν είναι για να προστατεύονται οι όσοι ε, παραβιάζουν τον νόμο, αλλά για να προστατεύονται οι πολίτες. Εδώ δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θώρακα που να είναι τόσο, μια πανοπλία που να είναι τόσο ε, δύσκολη στην αντιμετώπιση του και να προστατεύονται στο τέλος όσοι παραβαίνουν τον νόμο αντί να προστατεύονται οι πολίτες στα δικαιώματά τους ε, όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Και συμφωνούμε και επ' αυτού επίσης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Σμιτ και γι' αυτό, ότι οι διαδικασίες για την διαβίβαση και ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς οι διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κάποιες παρεκκλήσεις όσον αφορά την πρόταση με επιχειρήματα για παράδειγμα να διασφαλιστούν και να ε, υπάρχουν τα δικαιώματα των κρατών μελών να παρέχουν ή να μην παρέχουν αυτά τα στοιχεία και να μπορούν να αρνηθούν κιόλα και ρητά ή και σιωπηρά και να μην απαντούν μέσα σε ευλογές προθεσμίες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι χίλιες φορές πιο λειτουργικό θα είναι να έχουμε μια συγκεκριμένη προθεσμία για την ε, αποδοχή αυτών των στοιχείων. Και θα έχει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρνηθεί. Η, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κράτος μέλος θα έχει διορθώνει ο μιλητής το δικαίωμα να αρνηθεί. Και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να το δούμε αυτό, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Πρέπει να είναι ε, χρήσιμη η προθεσμία, να είναι αποτελεσματικού χαρακτήρα και μέσα στο ε, δικαίωμα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπίζει τα συμφέροντά της που είναι τα συμφέροντα όλων μας ε, φυσικά. Για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει δεν επικεντρώνονται αυτά τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι αυτά μπορούν να δημιουργούν δυσκολίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία που είχα είναι ακριβώς τα αντίθετα. Αυτή τη στιγμή ο κατακαιρματισμός στοιχείων είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί προβλήματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση απατών. Η συγκέντρωση και συλλογή αυτών των στοιχείων είναι προφανές ότι ε, ποτέ δεν θα έχουμε 100% αποτελεσματικότητα ευθύς εξ αρχής αλλά σταδιακά βήμα προς βήμα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα δίνουν τη δυνατότητα μέσα σε αποτελεσματικό εύλογο χρονικό διάστημα μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε ε, τέτοια συμβάντα. Θέλω να ευχαριστήσω και για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποτέ δεν ήμουν τελωνιακό εγώ κατά τη διάρκεια της ζωή μου, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι οι τελωνιακοί επίσης σε, σε όλες τις χώρες μας είναι οι πρώτοι, είναι οι πρώτες ε, που δημιουργήθηκαν. Οι κατηγορίες υπαλλήλων συλλογή εσόδων, φορολογικών εσόδων και τελωνιακοί υπάλληλοι στην πρώτη γραμμή των δράσεων αυτών. Έχω μεγάλο λοιπόν σεβασμό για, τις, ε, ε, για αυτή την πηγή εσόδων αλλά πρέπει επίσης να πω ότι έχουμε και, έχω εξίσου ε, σεβασμό για τους καταναλωτές και πρέπει και αυτοί φυσικά να προστατεύονται. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ε, συντάχθηκε και λειτουργήσε αυτή η έκθεση έτσι. Αν ήταν απλώς μια έκθεση για την ε, συλλογή σόδων, ε, τότε θα είμαστε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί. Βρισκόμαστε στη δική μας Επιτροπή για αυτή την πτυχή για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική σας δευτερολογία. Σίγουρα έχει γίνει πολύ και σκληρή δουλειά. Προθεσμή για την κατάθεση τροπολογιών, Τετάρτη λίγη, στις 12 το μεσημέρι. Λυπούμε, είναι πολύ σύντομο το χρονοδιάγραμμα, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε εξετάσει το έγγραφο ήδη. 3 Μαρτίου λοιπόν θα γίνει εξέταση των τροπολογιών στη συνεδρίασή μας και θα ψηφίσουμε στις 18 Μαρτίου. Ελπίζουμε, νομίζω έχουμε ήδη κλείσει αν θέλετε μια χρονοθυρίδα στην Ολομέλη για την ψηφοφορία, αλλά θα δούμε κατά πόσον θέλει να ε, συζητήσει το θέμα αυτό η Ελληνική Προεδρία. Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δύσκολα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα δούμε όμως πάντως αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να συμφωνείτε με αυτό. Περιμένουμε λοιπόν τις ε, τροπολογίες σας. 3 Μαρτίου θα τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε για πρώτη φορά εκπρόσωπος και φυσικά με τα χαρά να σας ξαναδούμε εδώ για να μας πείτε την άποψή σας για τις τροπολογίες. Έχουμε πέντε λεπτά παραπάνω στη διάθεσή μας από ό,τι είχαμε υπολογίσει γιατί προχωρήσαμε γρήγορα αλλά επειδή είναι εδώ ο κύριος Μάγερ μπορούμε να περάσουμε στο πακέτο ταξιδιωτικά μάλλον πακέτα. Υπάρχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Έχουν έρθει. Δεν ξέρω ακριβώς. Είναι έξω. Οπότε να τους δώσουμε ένα λεπτό για να έλθουν στην αίθουσα και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα καθυστερήσω λίγο να μπορέσουν να μπουν και να ακούσουν και τα σοφά λόγια του εισηγήτου. Πέντε λεπτά είπατε. Μάλιστα, άρα να καθυστερήσουμε λίγο, ώστε όλοι να είναι εδώ. Εντάξει. All right. Τέσσερις ακριβώς ε, θέλει ο σύντης μας να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, διακόπτουν πολύ σύντομα. Να έρθει και ο βοηθός ε, του βουλευτή, να έρθουν και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν. Μικρό διάλειμμα λοιπόν. Κυρίε και κύριοι, είναι ακριβώς τέσσερι η ώρα. Α αρχίσουμε λοιπόν. Υπενθυμίζω ότι είναι απολύτω ενδεικτικέ οι χρονοθυρίδε. Καμιά φορά λοιπόν αντί να καθυστερούμε μπορεί και να ε, τρέχουμε λίγο περισσότερο. Γενικά πάντως μας αρέσει να κρατάμε το χρονοδιάγραμμα της ε, ημερησίας διαταξής. Παρ' όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Μάιερ, καλώς ήρθατε. Καθώς και οι διάφορες και διάφοροι σκιώδεις συζητητές, οι αναπληρωματικοί τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω τον κύριο Κώστα Πέτρο, νομίζουμε ότι είπε ο πρόεδρος, και ο κύριος Ματιού. Θα μιλήσει ο κύριος Ματιού. Καλά. Ε, λοιπόν, καλώς ήρθατε και στο, στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες πριν από την αυριανή ψηφοφορία. Έχουμε 16 συνολικά. Θα δώσω τον λόγο στον ίδιο τον εισηγητή για να παρουσιάσει το αποτέλεσμα αυτό της εργασίας του και θα ακούσουμε μετά και από τους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Σμίτ αντικαθιστά τον κύριο Χέλβικ και άλλοι ευρωβουλευτές παρούσες ή παρόντες και έτσι χωρίς ε, περισσότερα λόγια από μέρους μου κύριε Μάγερ να σας δώσω το λόγο για να μας πείτε σχετικά με τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε συνολικά 435 τροπολογίες. Συν 100 τροπολογίες από την Επιτροπή Μεταφορών μαζί με τους ε, σκιώδους ηγητές καταλήξαμε σε 16 συμβαστικές τροπολογίες. Σε 5 συνολικά συνεδριάσεις με τους σκιώδους ηγητές. Ήδη λέγω από τώρα ότι αυτές οι συζητήσεις ήταν πολύ καρποφόρες και γόνιμες. Ιδίω δε η τελευταία συνεδρίαση με συμμετοχή των παρουσών και παρόντων συναδέλφων κατέσε δυνατό να καταλήξουμε σε συμβιβασμού στα πιο σημαντικά σημεία. Και θα αρχίσω με την πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό λοιπόν το click-through, το αφήνουμε εκτός του πεδίου εφαρμογή. Click-through που πάει να πει ότι ο ορισμός των ε, ταξιδιωτικών πακέτων, διότι για ένα συνολικό ολόκληρο ταξίδι δηλαδή, χρειαζόμαστε όλα τα δεδομένα, ενώ για ταξίδια που γίνονται, που κρίνονται δηλαδή κατά τμήματα, πρέπει ε, να υπάρχουν και λιγότερα. Για παράδειγμα, αν τώρα έχετε κλείσει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Παρίσι, μπορούν να σας προτείνουν και το τρένο για το Παρίσι. Δηλαδή καθαρά η διαφήμιση, αν σας πει κανείς, Μαγιόρκα από 1η μέχρι 7η Ιουλίου. Εκεί δεν εντοπίζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν ταυτοποιείται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν μπορεί κανεί να κάνει διαφήμιση τέτοια. Αυτή τη στιγμή όμω μπουν μέσα και δεδομένα του προσώπου, δηλαδή όνομα, ε, ημερομηνία γεννήσεω ή άλλα προσωπικά δεδομένα, αριθμό διαβατηρίου ή επιστοτική κάρτα κλπ. Οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, τότε δεν πρόκειται πλέον για διαφήμιση, αλλά για ταξίδι ενός από τα δυο είδη. Αυτό είναι και, το πιο, πιο σημαντική διαφορά. Ήδη μιλήσαμε με την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν εξακολουθεί να μην ενθουσιάζεται από τις ρυθμίσεις που προτείνω εμείς, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατό όταν κάποιος κλείνει ένα αεροπορικό ταξίδι ή ένα σιδηροδρομικό ταξίδι να μπορούν να γίνονται προσφορές εποφελία του καταναλωτού, να μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει μου αρέσει το τάδε ξενοδοχείο ε, ή όχι, χωρίς να χρειάζεται ο ίδιος να ψάχνει στο διαδίκτυο για να τα βρει. Όμως, ως δεδομένα επιτρέπεται να διαβάζονται μοναχά προορισμός του ταξιδιού και ε, ημερομηνίε. Όχι κανένα προσωπικό δεδομένο. Τώρα, δεν περιλαμβάνονται τα ευκαιριακά ε, ταξίδια που είναι συνολικά κλεισμένα, ενώ περιλαμβάνονται επιχειρηματικά ταξίδια εφόσον γίνεται η κράτηση μέσα στα πλαίσια μιας σύμβασης πλαισίου. Και σημειώστε ότι οι χώρες μέλη μπορούν να υπερβούν το πεδίο εφαρμογή της οδηγία με το ε, δίκαιο. Περιλάβαμε και ε, μια παράθεση από την Οδηγία Προστασίας του Καταναλωτού με σύστημα copy-paste, δηλαδή αυτούσια, ώστε να έχουμε ε, πραγματικά ακριβώς ίδιους, ίδιες διατάξεις. Τώρα, το άλλο θέμα είναι οι τροποποιήσεις των τιμών. Αυτό μόνο όταν δεν είναι κόστος του οργανωτή, αλλά εξωτερικά κόστη τα οποία αυξάνουν, για παράδειγμα, ε, τιμή της βενζίνης. Και εφόσον είναι παραπάνω από 3%. Από την άλλη μεριά, εάν υπερβαίνουν το 8%, τότε ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμιά επιβάρυνση. Έχει το δικαίωμα να λάβει ε, άλλη προσφορά σε σχέση με το αρχικό του ταξίδι και το ίδιο για αλλαγές οι οποίες ήδη έχουν, για τις οποίες έχουν ήδη γίνει ε, κρατήσεις. Όλα τα κόστη και όλα τα παρεμφερή κόστη θα πρέπει να επιστραφούν στην περίπτωση αυτή από τον οργανωτή. Τέταρτο, κατάλημα σε περίπτωση απρόβλεπτων ε, γεγονότων. Το ίδιο όπως για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρείων που και εκεί μετά από μακρότατες ε, συζητήσεις καταλήξαμε σε συμβασμό. Τον ίδιο συμβασμό νομίζω μπορούμε για λόγους διαφάνειας να υιοθετήσουμε και εδώ. Αυτό σημαίνει μέχρι πέντε διανυκτερεύσεις με maximum κόστος ανανύχτα 125 ευρώ. Εδώ υπάρχει βέβαια μια διαφορά ανάμεσα σε ένα καθαρό αεροπορικό ταξίδι και σε ένα συνολικό ταξίδι. Ο οργανωτής στη δική μας περίπτωση έχει τη δυνατότητα να οργανώσει πρώτο το κατάλημα και να το προσφέρει και αυτό του δίνει και τη δυνατότητα βεβαίως να μπορέσει να παραμείνει και κάτω από το όριο των 125 ευρώ. Θα πρέπει όμως να διατηρήσει, να λάβει υπόψη του τουλάχιστον την κατηγορία ξενοδοχείου που είχε κρατηθεί στην αρχή. Ή μπορεί να πει ότι παραμένει στο ίδιο ξενοδοχείο και δεν χρειάζεται ο ταξιδιώτης δηλαδή που καθυστερεί η πτήση του να μετακινηθεί από το ξενοδοχείο. Πέμπτο, παρεμπίπτουσες υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα μόνο του συνολικού ταξιδιού εφόσον προσφέρονται στους ταξιδιώτες εκείνους και εφόσον αυτές φτάνουν μέχρι το 25% του συνολικού κόστους. Για παράδειγμα μεταφορά γεύματα, καθαρισμός κλπ. που δεν είναι τμήματα του συνολικού ταξιδιού. Και είναι σημαντικό αυτό εάν μιλούμε για παράδειγμα για παραμονή σε ξενοδοχείο. Έκτο, σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας. Εκεί κάνουμε διάκριση ανάμεσα στον οργανωτή του ταξιδιού γιατί ο, ο που προσφέρει ταξίδι αλλά ανατμήματα είναι ο, για το κάθε τμήμα υπεύθυνο αυτός που το έχει οργανώσει. Και έβδομο, αλλαγές για την αντικειμενική ευθύνη των παρόχων ή των εμπόρων επεξεργαστήκαμε ένα συμβασμό που τα καλύπτει αυτά και δίνει στις χώρες μέλη τη δυνατότητα να καθορίσουν ορισμούς. Αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή, διότι υπάρχουν διάφορες χώρες μέλη που γνωρίζουν διαφορετικά είδη ευθύνη. Και αυτό είναι το μόνο άρθρο το οποίο επισέρχεται σε θέματα εναρμόνισης προς το συμφέρον της ενιαίας αγοράς και γι' αυτό εγώ σας παρακαλώ να το υποστηρίξετε όπως και την προσέγγιση που προτείνω εγώ, που πάλι ακολουθεί τις ρυθμίσεις της Οδηγίας Προστασίας Κατανολισμού. δηλαδή καταρχήν εναρμόνιση, αλλά με δυνατότητα εξαιρέσεων. Και αρχικά η Γαλλία, ο κ. Ζουβά, κατέθεσε τροπολογίες, αλλά και άλλες χώρες μέλη απεδείχθη ότι έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις και εφόσον αυτές οι διαφορετικές ρυθμίσεις εξυπηρετούν καλύτερα τους καταναλωτές, τότε μπορούν να τις διατηρήσουν οι χώρες μέλη. Αυτά είναι τα βασικά, μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα. Ούτως ή άλλως εμείς με τους συζητητές τα έχουμε συζητήσει επί ώρες. Αλλά θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές και εισηγήτρες για τη συνεργασία. Στην τελευταία συνεδρίαση των ε, σκιωδών εισηγητών, εγώ απέσυρα μία τροπολογία για το δικαίωμα ανακρίσεως. Διότι όταν κανείς κάνει τις κρατήσεις επιγραμμικά, έχει το δικαίωμα ανακρίσεως. Το διαδίκτυο, στο διαδίκτυο μάλλον, προσφεύγουν όλο και περισσότεροι. Και η οδηγία μας Μέχρι τώρα βεβαίω δεν λάμβανε υπόψη το διαδίκτυο, διότι όταν είχε τεθεί σε εφαρμογή δεν υπήρχε καν το διαδίκτυο. Όμως υπάρχουν τόσο πολλές διαφορές, για παράδειγμα και πτήσει στι οποίε ε, γίνονται κρατήσει για ε, περαιτέρω μετακινήσεις κλπ, ώστε απεφάσισα εν τέλει να το Παραμένει βέβαια το ίδιο της ε, Επιτροπής Μεταφορών. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια. Αυτά ε, καταρχήν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μας ε, ενημερώσατε, αλλά και για τη σκληρή δουλειά σας. Ξέρω πως κάνατε πολλές συνεδριάσεις για να μπορέσετε να συντάξετε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις των άλλων πολιτικών ομάδων, να δούμε πού έχει φτάσει η πρόοδος και θα αρχίσουμε με τον Αντιπρόεδρο Σέργιο Κονφεράτη, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Έχεις το λόγο, Σέργιο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους συναδέλφους τους σκιώδεις εισηγητές για την μεγάλη διαθεσιμότητα που έδειξαν στη διάρκεια της συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, αντικειμενικά ήταν δύσκολο το έργο μας, γιατί ξεκινάμε από ρυθμίσεις που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και άρα η εναρμόνισή τους είναι ένας στόχος ε, τον οποίο μπορούμε εύκολα να συμμεριστούμε, αλλά δύσκολα να επιτύχουμε. Έπειτα θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι και από την τεχνική ε, πλευρά το θέμα που μας απασχόλησε είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στους χρήστες και τους διαχειριστές της υπηρεσίας, δηλαδή τους εκείνους που προσφέρουν την υπηρεσία αλλά και εκείνους που στην ουσία το χειρίζονται στη συνέχεια. Παρά αυτή τη δυσκολία, νομίζω ότι η καλή θέληση που δείξαμε όλοι μας επέτρεψε να φτάσουμε σε κάποιες συμβαστικές που είναι σημαντικές και που είναι αυτές που τώρα μας παρουσίασε ο συνάδελφος Σμάγερ. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω μια συγκεκριμένη πτυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ορισμένες από αυτές τις συμβαστικές προτάσεις να επιβεβαιωθεί εκ νέου η βούληση των κρατών μελών να ενισχύσουν την προστασία του καταναλωτή, που είναι εξάλλου και ο στόχος της Επιτροπής μας και είναι πολύ καλό ότι, έχουμε, ότι, θα, ότι θα προτείνουμε λύσεις συναρμονισμένες εκεί όπου αυτό είναι δυνατόν. Αλλά δίνεται και κάποιο χώρο, κάποιο περιθώριο για προσθήκε από τα κρατημέλη, ώστε τα κρατημέλη δηλαδή να έχουν, αν το επιθυμούν, τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν ταξίδια κάτω των 24 ωρών ή να συμπεριλάβουν τις ενώσεις ε, που διοργανώνουν ταξίδια στην, ε, στην εφαρμογης εφαρμογή Όσον αφορά τώρα τι λύσει, η συμβαστική λύση που βρήκαμε είναι δεσμευτική. Κάναμε ένα βήμα μπροστά, νομίζω σημαντικό προ τη σωστή κατεύθυνση. Και θα ήθελα να πω στον εισηγητή, όπω και στου υπόλοιπου συνάδελφου, ότι αν με βάση τις πιθανές παρατηρήσεις της Επιτροπής ή με βάση τις παρατηρήσεις που έκανε η Επιτροπή Μεταφορών. Αν λοιπόν θεωρηθεί απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο του ορισμού όσον αφορά εμένα και τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, υπάρχει διάθεση να ξανασυζητήσουμε τα όσα ε, κάναμε μαζί. Είναι μια σημαντική πρόοδος, την οποία εκτίμησα εάν υπάρχει βούληση ή ενδιαφέρον ή και ανάγκη να ξανά κάνουμε ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας, από πλευράς μου είμαι διαθέσιμος να το ξανασυζητήσουμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένο για τις συμβιβαστικές για τα άρθρα 8 και 9 που εγγυώνται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη σύμβαση χωρίς τη συγκατάθεση του ταξιδιώτη. Και αυτό διότι προτιθέμεθα να ψηφίσουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να συζητηθεί με τους φυσικούς μας συνομιλητές, δηλαδή τη Γενική Κομισιόν και το Συμβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό να είναι πολύ ξεκάθαροι οι ορισμοί και να αιτιολογείται το γιατί θέλουμε να προστατέψουμε τον καταναλωτή. Και γι' αυτό και η δουλειά αυτή που κάνουμε ε, είναι πολύ δεσμευτική και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, οι θέσεις μας για κάποια πράγματα. Τώρα, ένα ακόμη θέμα Μάλλον κάποια άλλα θέματα δεν ε, ήταν αντικείμενα ε, συμβαστικών γιατί είναι υποσυζήτηση τροπολογία. Θα δούμε στη συνέχεια ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορία για αυτές τις ε, τροπολογίες. Είναι προφανές ότι η λύση που θα υιοθετηθεί κυρίως για ορισμένε από αυτές θα δώσει ένα ψηλό, μια, μάλλον μια ψηλότερο ή χαμηλότερο προφίλ ανάλογα με την πρόταση που θα εγκριθεί τελικά και ε, βέβαια ε, σε συνδυασμό με συμβαστικές προτάσεις. Και εδώ βέβαια θα εξαρτηθεί από τη σοφία της Ολομέλης, όπως έλεγε και ο ε, εισηγητής, να λάβει υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής μας, αλλά και τις προτάσεις που έκανε η Επιτροπή Μεταφορών, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις και οι πιο καλοί συνδυασμοί. Αυτό το πνεύμα λοιπόν, με το οποίο συζητήσαμε τις τροπολογίες μέχρι τώρα, θα πρέπει να δούμε και τη συζήτηση συζήτηση στην Ολομέλεια. Γιατί ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα στους χρήστες, το πρέπει να γίνει. Είχαμε μια διαρκή, διαρκή, σημείο αναφορά στην οδηγία περί καταναλωτών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πω ότι αυτή εδώ είναι μια καλή βάση για να προσπαθήσουμε μετά στη συνέχεια να προσθέσουμε ε, ε τους, ε, τα επόμενα λιθάρια για την οικοδόμηση του συνόλου ε, του κτίσματος. Σε ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία και να επαναλάβω ότι είμαι διαθέσιμος μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια να δούμε αν υπάρχει κάτι ακόμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ή άλλη καινοτομία. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέλβικ, ε, ε, μάλλον συγγνώμη, η κυρία Σπέκ, η οποία αντικαθιστά τον κύριο Χέλβικ. Σμιτ, με συγχωρείτε, ο κύριος Σμιτ. Ε, από ό,τι φαίνεται έχω αναλάβει ε, να εκπροσωπώ όλους τους φιλελεύθερους απόψε, λυπούμε γι' αυτό. Ο κύριος Χέλβικ ήθελε να σας ζητήσει συγγνώμη που δεν είναι σήμερα εδώ καταρχήν. Ε, καλωσορίζει τις συμβιβαστικές προτάσεις που έχουν ε, καταρτιστεί και ευχαριστεί τον εισηγητή και τους υπόλοιπους σκιώδεις για τη σκληρή δουλειά και την ευελιξία τους που μας επέτρεψε να συμφωνήσουμε σε αυτές τις συμβαστικές. Ο κύριος Χέλβικ μπορεί να υποστηρίξει τις περισσότερες τροπολογίες που αποσαφηνίζουν διάφορες διατάξεις της προτινόμενης οδηγίας. Εμείς η ομάδα ALDE έχουμε κάποια σημεία διαφωνίας, για παράδειγμα για το εκτιμώντας 17 όσον αφορά το ελάχιστο τμήμα και τις υπηρεσίες που είναι κομμάτι του πακέτου. Τώρα το πακέτο προτείνει 25% του συνόλου του πακέτου, για μας όμως είναι πολύ χαμηλό αυτό και Πιστεύουμε πως ε, θα διεύρυνε υπερβολικά το πεδίο τη οδηγίες, πράγμα που θα επηρέαζε τους μικρούς ε, φορείς στον τομέα. Ο κύριος Σέλβικ προτείνει το 40% που είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του πακέτου. Τώρα, συμβιβαστική 8 για την αιτιολογική σκέψη 40 μας ανησυχεί ότι το, άρθρο 8 της οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή θα ίσχυε εδώ και ε, επίσης θα πρέπει και αναφέρονται και οι επίσημες απαιτήσεις για τις εξαποστάσεως ε, συνάψεις, συμβάσεις, οι οποίες όμως καλύπτονται ήδη στο άρθρο 4 της παρούσας ε, οδηγίας, οπότε μπορεί να υπάρχει επικάλυψη. Αυτά, εκτός από ορισμένα μικρά σημεία που έχουν ήδη αναφερθεί, ο κύριος Σέλβεκ πιστεύει ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ θετική γιατί θα αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών, και ε, γιατί έτσι θα χαίρουν περισσότερη συνομικής βεβαιότητας. Σας ευχαριστώ. Και με χαρά σας βλέπουμε να αντιπροσωπεύετε εδώ όλους τους φιλελευθέρους. Το κάνετε με τόση πολύ ικανότητα που ε, τους αναπληρώνετε όλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή και ε, τις σκιώδεις εισηγητές. Ε, ε, δοθέτως και του περιορισμένου χρόνου, μεγάλη δηλαδή πίεση χρόνου που είχαμε, Καταφέραμε ωστόσο πολλά πράγματα. Υπάρχουν βέβαια ακόμα ορισμένα αμφισβητούμενα πράγματα όπως οι βοηθητικές υπηρεσίες που αναφέρατε πριν, ιδίως εκεί δεν περιλαμβάνεται ρητά το ταξίδι, travel δηλαδή, χρειάστηκε να ψηφίσουμε επίσης αν τα επιχειρηματικά ταξίδια θα μπουν στην οδηγία αυτή. Εγώ εξακολουθώ να μην είμαι πεπισμένη ότι θα, έπρεπε, ότι θα πρέπει να υπαχθούν εδώ. Και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα υπαναχωρήσεως οι προτάσεις σας με τις 24 ώρες και μόνο επιγραμμικά θα τα δεχόμουν. Αλλά οι προτάσεις που κάνει η Επιτροπή Μεταφορών μου φαίνεται αδύνατο να τις υποστηρίξω. Έχω να τονίσω ένα ακόμη πράγμα, σημαντικό για μένα. Όταν μιλούμε για όλο αυτό το πακέτο, είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι οι καταναλωτές δεν είναι όλοι ίδιοι, ούτε ίσοι, ούτε έχουν τις ίδιες επιθυμίες. Έχω την αντίληψη ότι ορισμένοι εδώ στην Επιτροπή βλέπουν μόνο ένα είδος καταναλωτού. Ενώ υπάρχουν διάφοροι τύποι καταναλωτών, για παράδειγμα ορισμένοι οι οποίοι επιθυμούν μοναχά κάποιες υπηρεσίες. Και καλά έκανε ο κ. Μάιερ και λέει ναι, έχουμε τα οργανωμένα ταξίδια, έχουμε τα άλλα που λέγονται συνδεδεσμένοι ε, διακανονισμοί και άλλοι ξεχωριστών υπηρεσιών που δεν συνδέονται με κάποιο σκοπό. Και εφόσον, αν βάλαμε μάλλον στην οδηγία, αν βάζαμε στην οδηγία αυτή, αυτές τις υπηρεσίες, τότε ε, θα χάνονταν και δεν ε, θα εξυπηρετούσαμε τους καταναλωτές. Δεν μπορεί λοιπόν ε, αυτό να είναι το νόημα της οδηγίας, διότι βλέπουμε όλο και περισσότερες νέους και νέους ανθρώπους που δεν θέλουν οργανωμένα ταξίδια, αλλά επιλεκτικά ορισμένες υπηρεσίες. Χαίρομαι λοιπόν που κάναμε τελικά το βήμα αυτό. Φοβόμουν στην αρχή ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Καταφέραμε όμως να κάνουμε καλά τον διαχωρισμό και σε ό,τι αφορά τώρα τα επιχειρηματικά ταξίδια και τις βοηθητικές υπηρεσίες, εκεί βέβαια τελικά θα χρειαστεί να ψηφίσουμε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μακ Λάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους συναδέλφους και για τη συζήτηση που είχαμε. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα, αλλά νομίζω ότι είναι καλές οι συμβαστικές προτάσεις στις οποίες καταλήξαμε σε ό,τι αφορά το πακέτο, τη συνδεδεμένα, τα συνδεδεμένα ταξίδια ε, linked travel. Νομίζω ο ορισμός είναι σαφής. Είναι σημαντικό να είναι σαφής η οδηγία και για τις επιχειρήσεις και για τους ε, πολίτες, πελάτες. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να περιλαμβάνει το πακέτο και το στοιχείο για τους, ε, ένα στοιχείο τους επιβάτες, ε, αλλά δεν το περιλαμβάνει τέλος πάντων όπως ορίζει το, το πακέτο όμως ε, είναι, με ικανοποιεί. Και σε ό,τι αφορά την 24ωρη αυτή περίοδο είναι σαφές και για το ταξιδιωτικό πακέτο και το, τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, το συνδεδεμένο ταξίδι. Είναι σαφές αυτό. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ε, που θέλω να αναφέρω και στον εισηγητή και στους σκιώδεις. Η μία αφορά το Linked Travel Arrangements, προσωρινά δεδομένα ε, και η μεταφορά των προσωπικών αυτών δεδομένων σε σχέση με τους δεκανούς που ισχύουν, χρόνος ε, και προορισμοί Ουσιαστικά εκεί βασίζονται και οι επιβάτες για την προστασία τους. Το να μην είναι λοιπόν ένα στοιχείο που θα πρέπει να μεταφέρεται, αυτό ενδέχεται να σημάνει ότι οι επιβάτες που βασίζονται σήμερα σε αυτό το νορισμό για τα μεταφορά δεδομένων δεν θα λαμβάνουν ε, το επίπεδο προστασίας που επιθυμούν και σίγουρα αυτό δεν είναι δική μας πρόθεση. Θα ήθελα λοιπόν να το αναθεωρήσουμε και να βάζουμε και τις ημερομηνίες ε, και τους προορισμούς για να μην μειώσουμε το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που ισχύει σήμερα και το οποίο αναφέρει και η Κομισιόν στην πρότασή της. Σε ό,τι αφορά το εκτιμώντας 17, έχουμε τις ίδιες επιφυλάξεις και με, όπως και η ομάδα ALDE για το ποσοστό των βοηθητικών υπηρεσιών. Δεν είμαι πεπισμένη ότι το 25% είναι αρκετά υψηλό ποσοστό, καλείται σημαντικό, significant παναλαμβάνω λοιπόν το αίτημά μου για 35%. Θα μπορούσαμε να το δούμε, ιδίω έχοντα ε, έχοντας υπόψη το 40% που πρότειναν ε, οι πράσινοι και οι άλντε. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να καταλήξουμε ε, σε ένα ενδιάμεσο ποσοστό. Χαίρομαι που λύθηκε το θέμα με το δικαίωμα επαναχώρησης για την 21 που θα προτιμήσω το αρχικό κείμενο της Κομισιόν σε ό,τι αφορά το κατάλημα, τη διαμονή. Δεν νομίζω ότι τηρούν τη διατάξεις του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών με, το, με την πρόταση ως έχει αυτή τη στιγμή. Ιδίω όταν δεν είναι ε, θέμα το οποίο υπόκειται στον έλεγχο των επιβατών το αν δηλαδή υπάρχει καθυστέρηση και θα πρέπει να τους παρασχεθεί κατάλημα. Επίσης, ο οργανωτής δεν θα πρέπει να έχει περισσότερες ε, δεσμεύσεις και περιορισμούς σε σχέση ε, με ένα τοξικό γραφείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 14, γίνεται χρήση της λέξης immediate, άμεσο, για την ε, αποζημίωση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Επίσης, να μην ε, ε, διευκολύνουμε τη μετανάστευση των επιχειρήσεων όταν μιλάμε για την έδρα, για την εγκατάσταση της επιχείρησης. Έχω και άλλες επιφυλάξεις για τις προτάσεις των σοσιαλιστών για τα άρθρα 8 και 9 όπως αυτές τις παρουσίασαν στην τελευταία συνεδρία επειδή συνεπάγονται μεγαλύτερο άχθος και για τις συγκεκριμένες συνθήκες και τις επιστροφές μειώσεις που προτείνονται. Καταλαβαίνω βέβαια ότι συμβιβασμός θα πει συμβιβασμός. Δηλαδή κάποιες φορές υπαναχωρούμε σε σχέση με κάποιες κόκκινες γραμμές που μπορεί να είχαμε. Ελπίζω να καταφέρουμε πάντως να συμβιβαστούμε πάνω στο ποσοστό, επαναλαμβάνω το αίτημά μου. Και για το δικαίωμα αναχώρηση είπαμε εντάξει, πρέπει να είναι ξεκάθαροι όροι πάντως και δεν θα πρέπει να προσελκύουμε ε, μάλλον δεν θα πρέπει να επηρεάζουμε τα επίπεδα προστασία των καναλωτών και να τα μειώνουμε. Good. Anybody Άλλος, κανείς θέλει να πάρει το λόγο, μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως είναι καλό που έχουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή αλλά και τους κοιόδης για τη δουλειά τους πάνω σε αυτό. Είμαι ευχαριστημένη που υπάρχει σύνδεση με το ταξίδι και άλλοι το είπαν, το γεγονός ότι δηλαδή που υποβοηθούμενο είναι περίεργο ε, αυτό συνδέεται με κάποιον που έχει κάποια αναπηρία και όχι με ε, τουριστικά πακέτα. Γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη αυτή η αποσαφήνιση. Οι τροπολογίε τώρα που διαπραγματεύτηκε ο κ. Κοφεράτη για τα άρθρα 8 και 9 είναι επίσης ευπρόσδεκτε και πιστεύω επίσης ότι τελικά προσπαθούμε να έχουμε μεγάλη σαφήνεια όσον αφορά την ευθύνη, γιατί αυτό είναι σημαντικό για την προστασία του καταναλωτή. Αύριο θα το ψηφίσουμε αυτό τώρα. Να ρωτήσω τον εισηγητή, ποια θα είναι η συνέχεια, θα υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Αν ναι, πότε και αν όχι, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσει αυτή η πρόταση και στο επόμενο κοινοβούλιο, στην θητεία. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος πως ο κύριος Μάιουρ θα μας τα πει όλα αυτά. Και βλέπω ότι ο Ντένις Διόγκ ήρθε. Α, ναι, μόλις έφτασε, εντάξει. Ναι, στο επόμενο. Μα γιατί σε έχω εδώ για σκιώδη και για τα τουριστικά πακέτα. Α, πολλά, πολλά σου πέσανε, μάλιστα. Ε, εντάξει, καλώς ήρθες πάντως. Άλλο άλλος κανείς θέλει να συμβάλλει. Πριν να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, να παρατηρήσω ότι έχουμε έναν εισηγητή από την Επιτροπή Μεταφορών που, συστήνει, που μάλλον συντάσσει χνομοδότηση. Ε, καλούμε τον κύριο Λιμπεράζη που είναι εισηγητής να έρθει και η κυρία Λίχτεμπεργκερ από τι νομικέ υποθέσει ε, συντάσσει γνωμοδότηση. Νομίζω όμω πω δεν είναι σήμερα εδώ, αλλά νομίζω ο κύριο Μάγερ έκανε ό,τι μπορούσε για να ε, εντάξει τι απόψει του σε αυτή την γνωμοδότηση. Ε, γι' αυτό για να δείξουμε ότι πάντοτε συνεργαζόμαστε αγαστά και με τις άλλες υπόλοιπε επιτροπές. Οπότε τότε να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Ματιά. Σας ευχαριστώ. Από πλευρά της Κομισιόν θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής μάλιστα για την ε, δουλειά τους ε, για τις συμβιβαστικές. Θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί ε, είναι πολύ καλές οι συμβαστικέ. Φυσικά θα πρέπει κάποιες από αυτές να τι μελετήσουμε πιο ενδελεχώ, αλλά για μας είναι σαφέ πω οι περισσότερε Είναι πολύ κοντά στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, πράγμα το οποίο καλωσορίζουμε. Επίσης καλωσορίζουμε το γεγονός ότι κάποιες διευκρινήσεις και βελτιώσεις ή προσαρμογές ε, στο κείμενο που το Υπάρχουν ωστόσο κάποια σημεία όπου βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες ε, ε, από, εκτροπές από την αρχική πρόταση της Κομισιόν και αυτές θέλουμε να σημειώσουμε. Ένα σημαντικό σημείο λοιπόν για μας ε, σχετίζεται με την τροπολογία υπαριθμών 4 που είναι ο ορισμός όσον αφορά το συνδυασμό διαφορετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών και διακανονισμών. Αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο. Αν δούμε τα κριτήρια που ορίζουν έναν συναφή ή συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ε, εδώ ορίζεται ένας πολύ στενός ε, ορισμός, απαιτείται δηλαδή ε, να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το όνομα του ταξιδιού ή οι επαφές, οι λεπτομέρειες της επαφής. Εδώ λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε σε τι ωφελεί αυτός ο ορισμός. Γιατί τελικά δεν θα έχουμε πολλούς συναφείς διακανονισμούς ή συνδεδεμένους ταξιδικούς διακανονισμούς, γιατί δεν θα μπορεί κανείς εύκολα να ε, ανταποκριθεί στις απαιτήσει αυτές και θα είναι αυτό μειονεκτικό για τον καταναλωτή. Επίσης πρόκειται για μια αλλαγή την οποία δεν είχαμε δει παλιότερα σε προηγούμενες συζητήσεις ε, στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών ας πούμε ή σε δηλώσεις που έγιναν προηγούμενα. Κάτι ακόμα αφορά την τροπολογία ε, υπαριθμών 7 η οποία έχει, αφορά την μορφή όπου η προσυμβατική ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται. Και εδώ προβλέπεται υποχρέωση για την προσυμβατική ενημέρωση μέσω, με, με κάποιο σταθερό μέσο. Εδώ η ανησυχία μας είναι πρακτικής μορφής, δηλαδή αν οι πρακτικές επιπτώσεις έχουν ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιγραμμικές συναλλαγές, δεν καταλαβαίνουμε πώς η υποχρέωση παροχής ενημέρωσης μέσα ε, ενός ε, μόνιμου μέσου, αν κάνει κανείς επιγραμμική κράτηση, α πούμε, ο διοργανωτής θα πρέπει να στείλει στον οποιοδήποτε καταναλωτή κάνει μια τέτοια κράτηση ένα email που περιλαμβάνει τις πληροφορίες της κράτησής του. Δεν βλέπουμε πώς στην πράξη μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω δηλαδή αν οι πρακτικές εφαρμογές έχουν ληφθεί υπόψη. Τρίτη σημείο είναι μια αλλαγή το θέμα της ευθύνης στην Κομισιόν είμαστε πεπισμένοι πως η λύση που προτείνουμε για την ευθύνη του διοργανωτή του οργανωτή είναι η καλύτερη λύση. Αλλά επίσης συνειδητοποιούμε πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. και ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η συμβιβαστική λύση. Τώρα προτείνεται να δοθεί κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι που μάλλον θα πρέπει να εξετάσουμε στην Επιτροπή καθώς που θα προχωρά αυτό το θέμα. Αυτά και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Good. Okay. Well, thank you very much. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να συνοψίσει με βάση και τα όσα άκουσε και αν έχει να μας πει τίποτα άλλο πριν από την αυριανή ψηφοφορία. και επίση να δούμε και ποια είναι τα επόμενα βήματα που προτείνετε την ερώτηση κύρια κυρίας Νομίζω στόχο έχουμε την Ολομέλεια του Μαρτίου. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι η ψηφοφορία θα πάει καλά αύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σας δώσω το λόγο τώρα για να μας πείτε εσείς τη γνώμη σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ παρόλα αυτά όλες και όλους για τις τοποθετήσεις σας. Το θετικό είναι ότι σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνεται συμφωνία. Οι περισσότερες τοποθετήσεις άλλωστε αυτό το νόημα είχαν, διότι αφενός θέλουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη εναρμόνιση γιατί έχουμε την ενία αγορά και θέλουμε οι δυνατόν όλοι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, από την άλλη μεριά οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών. Έχουμε λοιπόν σε ορισμένες από τις συμβαστικές τροπολογίες επιτύχει ακριβώς αυτό. Κοινά δικαιώματα και ταυτόχρονα δίνουμε κάποιο περιθώριο στις χώρες μέλη. Ή στα θέματα, για παράδειγμα, της ευθύνη, εάν δηλαδή θα είναι μόνος οργανωτής εκείνος ο οποίος θα έχει την ευθύνη, είτε ο διαμεσολαβητής για το δικό του μέρος της δουλειάς, είτε και οι δυο μαζί. Ε, η δική μας ρύθμιση είναι ο καθένας να φέρει την ευθύνη για το δικό του τμήμα. Οι χώρες μέλη όμως έχουν το δικαίωμα να δώσουν με τη σειρά τους στον καταναλωτή το δικαίωμα να στραφεί και κάτω των δύο. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία για τον καταναλωτή. Και γι' αυτό δεν είμαστε αντίθετοι αν θέλουν οι χώρες μέλη να προβλέψουν κάτι τέτοιο. Ο κ. Κοφεράτη άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Κύριε Σμιτ, για τον ε, για την ομάδα Άλντε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για την ε, τροπολογία 17, ε, για το 40% των βοηθητικών υπηρεσιών. Φτάνουμε όμως κοντά στις, ε, κυρίως στις ουσιώδεις υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι το 50% τουλάχιστον. Σε πολλές συζητήσεις βεβαίως τα είπαμε αυτά. Μπορούμε δηλαδή να διευκολύνουμε εδώ με την έννοια ότι δεν θα είναι οι ουσιώδεις υπηρεσίες τόσο το μεγαλύτερο μέρος ε, των δαπανών, αλλά ο σκοπός ταξιδιού. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να θέλει να πάει σε μια θεατρική παράσταση ή ε, να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Και το υπόλοιπο κόστος ταξιδιού να είναι πολύ υψηλότερο. Αν όμως το ποδόσφαιρο ή το θέατρο είναι ο βασικός σκοπός του ταξιδιού μου, έστω και αν είναι μόνο το 15% του συνόλου κόστους, θα πρέπει να είναι αυτό που θα παίξει το ρόλο. Άρα θα πρέπει να υπάρξει κάποιο συνδυασμό μεταξύ τιμή και σκοπού του ταξιδιού. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούμε του περισσότερους καταναλωτές. Έτσι νομίζω. Για την κυρία Ρούλε τώρα. Παρεμφερείς υπηρεσίες ή ε, ε, η πρόταση ήταν από 3% μέχρι 50%. Έτσι. Και με 435 τροπολογίες καταλαβαίνετε. 3% μου φάνηκε υπερβολικά λίγο, 5% μου φάνηκε υπερβολικά πολύ. Γι' αυτό καταλήξαμε τελικά στο 25% μέσα σε αυτή την παραδοσιακή ε, προσπάθεια, ευρωπαϊκή προσπάθεια συμβιβασμού. Τα επιχειρηματικά ταξίδια τώρα δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας μας εφόσον κρίνονται μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτου αξιδιού. Αν όμως ένας ελεύθερος επαγγελματίας, δικηγόρος, ε, ιατρός, κλείνει ένα τέτοιο ταξίδι, τότε υπάγεται στην προστασία του νομοθετήματος. Ούτε μπορεί να εκπέσει της προστασίας μόνο και μόνο επειδή ασκεί ένα επάγγελμα, όπως είπα ιατρός ή α, ε, μηχανικός ή κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε και εδώ λοιπόν να ειδούμε τα, τα, τα επαγγελματικά ταξίδια ξεχωριστά. Αν και βέβαια και ο επιχειρηματίας εφόσον κλείνει ιδιωτικό ταξίδι πρέπει να μπορεί να προστατεύεται. Για την κυρία Μακ Λάρκιν, ο ορισμός του οργανωμένου ταξιδιού μας απασχόλησε πολύ. Και τις 24 ώρες τις δεχτήκαμε όπως επιθυμούσατε εσείς. οι επιφυλάξει σχετικά με, τη διαβίβαση δεδομένων στου συνδεδεμένου ταξιδιωτικού ταξιδιωτικούς Κοιτάξτε, για την αρνητική οριοθέτηση. Ε, εάν θέλουμε να αφήσουμε στον ταξιδιώτη να έχει τη δυνατότητα δηλαδή να βλέπει τις διαφημίσει, και εγώ νομίζω ότι πρέπει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια πράγματα επιτρέπεται να διαβιβάζονται περαιτέρω με τα κλικ που κάνει στον υπολογιστή του ο ταξιδιώτη χωρί να προκύπτει δέσμευση γι' αυτόν. Αν δηλαδή διαβιβάζονται μοναχά ο προορισμός του ταξιδιού και το χρονικό πλαίσιο χωρίς προσωπικά δεδομένα, τότε πρόκειται διαφήμιση και δεν υπάγεται στην παρουσαδία. Αν θέλω να πάω μία εβδομάδα στη Μαγιόρκα στις αρχές Ιουλίου, 1η έως 7η Ιουλίου, και το μόνο που διαβιβάζεται είναι Μαγιόρκα και 1η έως 7η Εβδόμου. Κανένα δεν μπορεί να πει τώρα είναι ο κύριο Μιούλερ, είναι ο κύριο Μάγερ, είναι η κυρία Μακλάρκιν. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αναφορά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο ή άλλο προσωπικό δεδομένο. Αυτή είναι η απόλυτη προπόθεση. Από την άλλη μεριά, εάν κάτι παραπάνω διαβιβάζεται, τότε μπαίνουμε αμέσω στο οργανωμένο ταξίδι, όπω θέλετε πέστε το, αλλά γι' αυτό απαιτούνται και περισσότερα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να λέει εγώ Πέτερ Μάιερ επιθυμώ να μεταβώ στο τάδε μέρο, στο τάδε χρόνο και υπό αυτέ τι συνθήκε. Προσπάθεια λοιπόν οριοθετήσεω είναι αυτή που κάνουμε. Τώρα, αποζημίωση. Άμεση αποζημίωση, αμελητή αποζημίωση, πολλές ε, εκφράσεις χρησιμοποιήθηκαν. Αν πούμε άμεση αποζημίωση και βεβαίως η γλωσσομαθείς νομικοί θα μεταφράσουν ε, αναλόγως. Δηλαδή στην πραγματικότητα αποζημίωση χωρίς καμιά ιδιαίτερη καθυστέρηση. Δεν ανάγκη να είναι αυθημερών ούτε την επόμενη μέρα. Αλλά πάντως αποζημίωση χωρίς καθυστέρηση. Ε, πάλι αυτή είναι η συμβαστική λύση στην οποία καταλήξαμε. Λύση στην οποία καταλήξαμε. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα, όντως αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην ολομένη θα ψηφίσουμε τον Μάρτιο. Η ελληνική προεδρία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει, ούτε έχει και καμιά πιθανότητα στο πρώτο αυτό εξάμεινο να ολοκληρώσει το θέμα, γιατί και εμείς διακόπτουμε τις εργασίες μας στην ουσία από τα μέσα Απριλίου. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να προχωρήσουμε σε τριμερείς διαλόγους. Άρα εμείς εδώ καταλήγουμε στην πρώτη ανάγνωση και σύμφωνα με τους κανονισμούς μας το νέο κοινοβούλιο θα αναλάβει την σκητάλη από εκεί και πέρα. Αλλά από το σημείο αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεται από την αρχή. Έχουμε λοιπόν μια ασυνέχεια όπου και αν βρίσκεται μάλλον στην Γερμανική Βουλή ε, σημειώνει ο κ. Μάιερ Έχουμε την ασυνέχεια, δηλαδή όπου και έχει, φτάσει, και έχει ένα νομοθέτημα, με τη λήξη θητεία αναλαμβάνει από την αρχή το επόμενο κοινοβούλιο. Ενώ εδώ ευτυχώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει η συνέχεια. Τώρα, έχουμε πάρει υπόψη και τι ε, τροπολογίε Νομική Επιτροπή και Επιτροπή Μεταφορών, στο βαθμό που ήταν δυνατό. Με την Κομισιόν θα συζητήσουμε. Μέχρι τώρα βεβαίω έχουμε συζητήσει πολύ σύντομα μόνο για τον ορισμό των ε, συνδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών. Τώρα το άλλο, το διαρκές μέσον. Με την έννοια αυτή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email, ικανοποιεί τον ορισμό αυτό. Με κάποιο τρόπο πρέπει να λαμβάνει ο ταξιδιώτης κάποια πληροφορία για τα δικαιώματά του. Και στις σημερινές εποχές του email, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι και το πιο ταχύ αλλά και το πιο εύκολο και ενδεδειγμένο κατά τη γνώμη μου μέσο για να πληροφορηθεί ρητά ο καταναλωτής για τα δικαιώματά του. Τέλος μίλησε η Επιτροπή για την ευθύνη. Νομίζω ότι είναι καλή η λύση που δώσαμε, δηλαδή για το, για το οργανωμένο ταξίδι ευθύνεται συνολικά ο διοργανωτής. Για, τα, για τους συνδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ευθύνεται ο καθένας για το κομμάτι του. Αν όμως υπάρχουν χώρες μέλη όπου οι συνήθειες είναι διαφορετικές, και επιτρέπουν στον καταναλωτή να στραφεί κατά περισσότερων προσώπων, γιατί όχι. Σημαίνει μεγαλύτερη προστασία για τον ίδιο. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Νομίζω ότι μετά από μια σύντομη συζήτηση θα μπορέσουμε αύριο να ψηφίσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Μάγερ που μας καθοδηγείτε με την πολύ σημαντική σας δουλειά σε αυτό το θέμα. Όπως είπατε, σαφείς ενδείξεις από πλευράς ελληνικής προεδρίας ε, δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμο το Συμβούλιο να συζητήσει μαζί μας αυτό το στάδιο. Η έκθεσή μας λοιπόν που ελπίζουμε να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια θα συμβάλλει και βέβαια ελπίζουμε να λάβει σοβαρά και το Συμβούλιο το θέμα αυτό. Οπότε πλέον θα περάσει στην Ιταλική Προεδρία που φαίνεται να έχει μεγάλες φιλοδοξίες και ελπίζουμε αυτοί να θελήσουν να προωθήσουν ε, το φάκελο. Πάντως εμείς ε, νομίζω ότι βελτιώσαμε σημαντικά την πρόταση και Πρώτα απ' όλα προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία και εργαζόμαστε σκληρά ώστε να έχουμε αρκετές πιθανότητες να το συζητήσουμε το Μάρτιο γιατί είναι σημαντική ε, πρόταση και για τους καταναλωτές και για πολλές επιχειρήσεις ε, που ε, ασχολούνται με τους πελάτες αυτούς, με τους καταναλωτές αυτούς. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε. Σας ευχαριστώ όλους και τώρα μπορούμε να περάσουμε αμέσως ε, στο τελευταίο για απόψε θέμα της μέρης διάταξης και συγκεκριμένα στη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Οικονομικών και Θεμάτων σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν, πρόταση κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με χρήση καρτών. Ο κύριος Μπίλαν είναι μας, ε, είναι εδώ. Κύριε Μπορίσοφ, μάλλον. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ. Τον κύριο... Κύριε Μάγερ, θα εσείς θα εκπροσωπήσετε τον κύριο Μπορίσοφ, μάλιστα. Η κυρία Βερνιό, σκληρά εργαζόμενη αντιπρόεδρος από την ομάδα σοσιαλιστών, Σμιτ εδώ για αυτή τη φορά είναι και σκιώδης ο ίδιος, δεν αντικαθιστά κάποιον άλλο. Ο κύριος Ντεγιόγκ είναι εδώ. Κυρία Βάιζεμπεκ, χαίρομαι που σας βλέπω. Θα μιλήσετε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, ωραία. Καλώς ήλθατε για μια ακόμη φορά. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπίλαν για να μας παρουσιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας υπενθυμίζω ότι θα ψηφίσουμε αύριο και για αυτή την γνωμοδότηση. Και όσοι δεν ήσασταν νωρίτερα, ε, να έχετε υπόψη ότι αύριο έχουμε μια αλλαγή στη ψηφοφορία, δηλαδή θα ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Μπίλαν και μετά την έκθεση Μάγερ. Ή ανάποδα τα είπα, κυρία Βερνιό. Όχι, σωστά τα είπα, μάλιστα. Συγγνώμη, πέθαλα να είμαι σίγουρος ότι θα είναι και η κυρία Βερνιό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπίλαν, συμβαστικές τροπολογίες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συνεδριάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους σκιώδες εισηγητές στο Στρασβούργο. Όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων ήταν παρόντες. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση, διότι λάβαμε μια σειρά από αποφάσεις ε, και εγκρίναμε πολλές συμβαστικέ προτάσεις, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Άρα οι πολιτικές ομάδες έχουν καταλήξει σε συμφωνία, βελτιώσαμε τις, ε, τους ορισμούς ό,τι αφορά τις πληρωμές ε, μέσω πιστοτικών χρηστικών καρτών, ε, την ορισμό των καρτών πληρωμών και αποφασίσαμε οι συντονιστές να υπογραμμίσουμε τη σημασία και της ελάχιστης εναρμόνισης αυτής της έννοιας. Αυτό τι σημαίνει ότι στο άρθρο της έκθεσης θέλουμε να γίνεται αναφορά στο εκτιμώντας 14, στην εντολική Σκέψη 14. Δηλαδή να ορίζονται πιο χαμηλές τραπεζικές ε, προμήθειες από αυτές που προβλέπει ο κανονισμός. Επίσης συμφωνήσαμε να υπάρξει συντόμευση των προθεσμιών εξέτασης ε, επειδή είναι πολύ ραγδαίες οι εξελίξεις στον τομέα αυτό, από 4 σε 2 έτη λοιπόν. Για να μην καθυστερούμε να ε, λάβουμε πόσο μας όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν. Δύο χρόνια λοιπόν μετά την έναρξη ισχύω του κανονισμού Άρα ουσιαστικά τέσσερα χρόνια από τη, από θα επανεξετάσουμε και θα αναθεωρήσουμε το πώς επηρεάζει οι διατάξεις αυτές τη λειτουργία της αγοράς. Θέλουμε η Κομισιό να προσέξει πολύ την αγορά αυτή, να δει τι εμπόδια ενδέχεται να προκύψουν υπάρχουν έμεσα κάποιες διατραπεζικές προμήθειες που πρέπει όλα αυτά να τα μελετήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 3 και 4, τις διατραπεζικές ε, προμήθειες και τις προθεσμίες, μετά από συζητήσεις καταλήξαμε στη διατήρηση των ε, κατώτατων ορίων της Κομισιόν. Υπήρξαν διαφωνίες, υπήρξαν διαφορές απόψεων. Τελικά όμως ε, οι περισσότερες πολιτικές ομάδες συμφώνησαν να παραμείνει η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σε ό,τι αφορά τις μεταβατικές περιόδους, θέλουμε να υπάρξει αναρμόνιση για τις εθνικές και διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Μελετήσαμε επίσης ε, το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός σταθερού συντελεστή για τις πολύ μικρές πληρωμές τα micropayments. Θέλαμε να βρεθεί μια λύση για αυτές τις πάρα πολύ μικρές πληρωμές, ώστε να καλύπτονται όλες οι χρεώσεις ε, επεξεργασίας. Δυστυχώς όμως φοβούμε ότι δεν ε, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να εξολογήσουμε τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια διάταξη. Αυτή τη σταθερή προμήθεια, αυτό το συντελεστή, το σταθερό, τον προτείνει ο κ. Δεν νομίζω όμως ότι συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες με την πρότασή του. Θα πρέπει λοιπόν ε, να τη σκεφτούμε. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να πετύχουμε το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή οι καταναλωτές να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν ε, κάρτες. Αυτό όμως δεν είναι δική μας πρόθεση. Εμείς θέλουμε οι καταναλωτές να επιλέγουν πάντοτε την καλύτερη λύση. Είναι και θέμα χώρας. Ποιος, συντελεστή θα χρησιμοποιείται για μια συναλλαγή στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Και τι είναι μια πολύ μικρή πληρωμή, micropayment. Άλλα, άλλα ε, ισχύουν στη Βουλγαρία, άλλα ισχύουν στη Σουηδία, για παράδειγμα. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα αυτό η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, πιστεύω, η ΕΚΟΝ δηλαδή, θα πρέπει να εγκύψει στο θέμα αυτό. Θα μπορούσα στις συμβιβαστικές μου προτάσεις να το συμπεριλάβω ε, το θέμα αυτό. Είμαι πάντως ε, ανοιχτός ε, στις προτάσεις των συναδέλφων. Αυτά είχα να πω. Αύριο ψηφίζουμε. Ελπίζω να εγκριθεί η γνωμοδότηση Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ε, τους κοιότητες εισηγητές και όλους όσους συμμετείχαν ε, στις εργασίες και βέβαια και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο και τη γραμματεία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε λοιπόν τις πολιτικές ομάδες. Κύριε Μάιερα, πρώτα, εξ ονόματος του ΕΛΚ, παρακαλώ. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. τι να πω, αν μου αρέσουν, αρέσουν, ότι αρέσουν και στον κύριο Μπόρισοφ. Θα ήθελα λοιπόν να πω, ευχαριστώ τον κύριο Μπίλαν, καθώς και τους υπολείπους για τη συνεργασία τους. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε θετικούς συμβασμούς και ως ο ηγητής του Λαϊκού Κόμματος υποστηρίζω τις συμβαστικές 1 και 2 για τον ορισμό των πιστοτικών και των χρεωστικών καρτών, την υπαριθμόν 3 για τον ορισμό της κάρτας πληρωμής όρου που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνώ ότι θα πρέπει να οριστεί ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια. Υποστηρίζω και την συμβαστική τροπολογία 4, δηλαδή σε δύο χρόνια μετά από τη θέση εφαρμογή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετική με την εφαρμογή. Ελπίζω ότι το χρονικό αυτό διάστημα θα είναι αρκετό για να παραγάγει αποτελέσματα ο κανονισμός και για τα interchange fees που ήταν το πιο προβληματικό θέμα συμφωνήσαμε σε ένα επίπεδο 0,2% για τις χρεωστικές και 0,3% για τις πιστοτικές κάρτες. Αυτές οι οροφές θα επιβληθούν σε όλες τις διαμεθοριακές πληρωμές με κάρτες μέσα σε, δύο, σε ένα χρόνο. Αυτό είναι το καλύτερο νομίζω για να μην ανησυχεί τους καταναλωτές. Εγώ υποστηρίζω και τις αρχικές προτάσεις της Γιόγκ για τις μικροπληρωμές, όπου οι χώρες μέλη μπορούν να επιβάλλουν ένα ελάχιστο τέλος για τέτοιες συναλλαγές που γίνονται με οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστοτική κάρτα. Εν τέλει θα ήθελα να σας επισημάνω την πρόταση του All Guards Rule που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να έχουν την ίδια κάρτα, το ίδιο τέλος συναλλαγής μάλλον, όμως τότε πιστοτικές και εμπορικές κάρτες θα πρέπει να έχουν μια, ένα ανώτατο όριο. Εκτός αυτού, οι καταναλωτές δεν θα έχουν και βεβαιότητα για το εάν η κάρτα τους θα γίνει αποδεκτή ή όχι. Το οποίο θα τους αποθαρρύνει να πληρώνουν με κάρτα και αυτό είναι αντίθετο βέβαια με το σκοπό του κανονισμού. Γι' αυτό και σας προσκαλώ να, να υποστηρίξετε τη δική μου τροπολογία υπαριθμών 80 που διαγράφει τον κανόνα on all cards. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ το λέω αυτό, ως Μάιερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ξεκάθαρα αυτά που μεταφέρατε διαστόματός σας από τον κύριο Μπορίσοφ. Κύριε Βερνιό, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν είχαμε και σημαντικά προβλήματα με αυτή τη γνωμοδότηση συνολικά. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον εισηγητή μας κύριο Μπίλαν, που ακολούθησε μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση, μας πρότεινε συμβιβασμού ε, που συνολικά έγιναν ε, δεχτεί θετικά από όλες τις πολιτικές ομάδες. Χαίρομαι ιδίως για τις τροπολογίες που έχουν ως στόχο την ε, διευκρίνηση ορισμών και απλούστευση της δομής του κειμένου και αφήνουν λίγο περισσότερο χρόνο ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τις διατάξεις του κειμένου. Χαίρομαι επίσης που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να μελετήσει την κατάσταση αυτών ε, των τριμερών συστημάτων. Ιδίω όταν βλέπουμε να υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις ε, συγκεκαλυμμένες προμήθειες και με όχι αμεληταία ποσά. Καλό επίσης συναδέλφους μου να στηρίξουν ορισμένες τροπολογίες της δικής μου πολιτικής ομάδας που νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν ε, πρόσθετη αξία για το κείμενο. Δηλαδή να μην περιοριστούμε σε τροποποιήσεις των όρων μεταξύ τραπεζών, αλλά να έχουμε μια πραγματική βελτίωση για τον καταναλωτή και για τον επιχειρηματία, τον έμπορο. Γι' αυτό θέλω την τροπολογία 79 να τη στηρίξετε. Η τροπολογία αυτή ε, προβλέπει η μείωση ε, των ε, διασυνοριακών προμηθειών ε, ε, να ε, μετακυλίονται στον καταναλωτή και τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με ενημέρωση του καταναλωτή για τις επιβαρύνσεις όλων των συστημάτων καρτών πληρωμών. 74, 75 και 87 τροπολογίες. Σύμφωνο την είναι έκθεση. Συνολικά θα ήθελα βέβαια να είναι λίγο πιο μεγάλη ευελιξία που θα είχαν στη διαθεσία τους τα κράτη-μέλη για να μπορούν να ορίζουν τα ανώτατα όρια μέσω των χρεωστικών πληρωμών για να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση που ισχύει στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Υπάρχει βέβαια και το διασυνοριακό εμπόριο. Είναι καλή δουλειά που έγινε. Θέλω να συγχαρώ όχι μόνο τον συγκεκριτή, όλου του σκιώδει, να συγχαρώ και αυτού Νομίζω εργαστήκαμε με ευρωπαϊκό πνεύμα που θα πρέπει να έχουν όλοι και σε άλλες επιτροπές. Όχι μόνο στη δική μας. Ευχαριστώ. Thank Uh... Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σμιτ. Um, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Μπίλαν γιατί νομίζω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά και μπορώ να υποστηρίξω όλες τις συμβιβαστικέ. Αλλά Πρέπει να πω αρχικά ότι μπορεί κανείς να νομίζει πως είναι πολύ εύκολη αυτή η νομοθεσία, αλλά δεν είναι για μένα. Εγώ ήμουν κατά εξ αρχής. Δεν είναι εύκολες, ε, εύκολη καιρή για φιλελεύθερους. Αλλά δεν είμαι υπέρ ενός ανώτατου όριου ως αρχή. Αυτό είναι λάθος, βασικά. Αλλά τώρα νομίζω πως κάτι πρέπει να κάνουμε ε, είχαμε και διάφορες συστάσεις από πλευράς του Κοινοβουλίου παλιότερα, αλλά πρέπει να ομολογήσω πως δεν τις είχα υπερψηφίσει. Ε, νόμιζα πως ε, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να προσαρμοστούν και να εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό και εντάξει μπορεί να είμαι και λίγο αγαθός λίγο αγαθός σαν φιλελεύθερος πάντως τώρα είμαι υπέρ αυτού εδώ και έχω ακούσει επικρίσεις γι' αυτά, αλλά δεν με πειράζει. Νομίζω πως είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι ε, μία μέση οδός πάντοτε είναι καλύτερη όταν ε, είναι μυστήριο το θέμα. Πάντως εδώ είναι αποδεκτά όλα αυτά και αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά λειτουργούσα ενιαία αγορά ε, πρέπει κάτι να κάνουμε για όλα αυτά. Ακόμα και οι Αμερικανοί κάναν κάτι για όλα αυτά. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Είναι σαν να λέει κανεί. εντάξει κάνω και το σταυρό μου, αλλά θα το κάνω. Τώρα για τις μικροπληρωμές. Κύριε Μπίλαν, το είπατε, είπατε ότι έχουμε αργήσει πολύ για όλα αυτά. Ελπίζω πως όχι όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και το συζητήσαμε στη συνάντησή μας στο Στρασβούργο. Νομίζω πως ο κύριος Ντεγιόγκ κάτι έχει καταφέρει εδώ, στη χώρα μου. Αυτές αυξάνονται με, με πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αν δεν μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε, δεν το, εντάξει, δεν το νομίζω πως... Δεν μ' αρέσει και πολύ. Όλοι θα πρέπει να έχουν και κάποια ψηλά στην τσέπη τους. Αλλά πάντως έτσι πάει το πράγμα. Όλο ένα και πιο πολλές μικροπληρωμές γίνονται για οτιδήποτε. Για μια σοκολάτα, για μια εφημερίδα, ό,τι να είναι. Και τι... Ελπίζω λοιπόν πως και εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε, να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία, γιατί σε άλλες συμβαστικές συμφωνώ, το ξέρετε. Κατά τα λοιπά σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά. Thank you for your clear exposition. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σαφήνειά σας και για την πολύ ρεαλιστική σας προσέγγιση. Κυρία Ρούλε, όχι. Ο κύριος Τζεγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή γιατί είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση σύσκεψη στο Στρασβούργο και μάλιστα η ομάδα μου πολύ ευχαρίστως στηρίζει τις προτάσεις του. Ανέφερα ένα θέμα το οποίο ε, είναι κάπως προβληματικό, όπως είπε και ο Όλε Σμιτ, γιατί είναι δύσκολος ο τομέας και υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα. Κάτι που ήθελα να ορίσουμε είναι το μακροπρόθεσμο συμφέρον του καταναλωτή να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν είτε μια κάρτα που εκδίδεται από αμερικανική εταιρεία, η Mastercard, η Visa ας πούμε, δεν είναι και τόσο πολλές οπότε μπορώ να τις αναφέρω, αλλά να έχουν και την επιλογή για μια ευρωπαϊκή κάρτα. Υπάρχουν μικρότερες κάρτες σε κάποιες χώρες μέλη όχι σε όλες τις χώρες πια, γιατί στις ε, κάτω χώρες το δικό μας εθνικό σύστημα αγοράστηκε από την ε, Mastercard, το μαέστρο που λεγόταν. Οπότε η επιλογή του καταναλωτή είναι πολύ πολύ μικρή. Πρέπει να βασιστούμε δηλαδή σε αυτό το σύστημα, ιδιαίτερα για τις μικρές πληρωμές, μικροπληρωμές όπως λέγονται. Από αυτής της ε, Βάσεις λοιπόν, πιστεύω πως ήταν απαραίτητο να το, προσέξουμε αυτό και ίσως και να μην ε, το ορίσουμε υπερβολικά, γιατί αρχικά είχα, μια, είχα καταθέσει μια τροπολογία ορίζοντας το ποσό που κανείς μπορεί να χρεώσει για μικροπληρωμή, για κάθε μάλλον μικροπληρωμή, αυτό δεν είναι πολύ δημοφιλεύς ε, βέβαια για τους μαγαζάτορες, ε, γιατί πρέπει κανείς και όλας να περιμένει και τα λοιπά. Κάναμε μια σχετική συζήτηση στους, ε, ανάμεσα στους κοιόδες και να πούμε αφήστε το στα κρατημέλη, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να γίνει, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και μικρότερες κάρτες, γιατί μακροπρόθεσμα είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών να έχουν μια επιλογή αλλά και προς το συμφέρον των ε, καταστηματαρχών να έχουν επιλογή ποια κάρτα δέχονται και ποια όχι. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο, ήδη είχαμε δύο ομάδες που το στηρίζουν και τουλάχιστον ε, αναφέρετε και τονίζετε το πρόβλημα για την ΕΚΟΝ. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε να συμφωνήσετε και για αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ όλους. Επικοδομητικές ιδέες και προτάσεις. Θέλει κάποιος άλλος να συμβάλλει στη συζήτηση, η κυρία Στάιλερ. Ναι. Γρήγορα, γρήγορα, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδης. Κατατέθησαν διάφορες τροπολογίες και με χαρά βλέπω ότι ο εισηγητής στηρίζει την προφορική με βάση την οποία τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εισάγουν δικά τους μέτρα Χαίρομαι που βλέπω να στηρίζεται αυτή η τροπολογία. Επίσης έγιναν δεκτές πολλές από τις δικές μου τροπολογίες και αυτό με ενθαρρύνει γιατί πιστεύω πως είναι περίπλοκο το θέμα και για πολύ κόσμο είναι ένας τομέας όπου όταν κανείς αρχίζει να μιλά για αλλαγές είναι κάτι που ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί πόσο πολύ τον επηρεάζει. Τώρα μόλις μιλήσαμε και είπαμε ότι είναι επιστοτικές κάρτες για το κόστος, για το πόσο σε χρεώνουν όταν τις χρησιμοποιείς κτλ. Τότε ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όντως τον ε, ε, αγγίζει άμεσα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Εμεί είμαστε επιτροπή που γνωμοδοτεί. Η ΕΚΟΝ είναι η αρμόδια από τι ουσίε. Πώ θα αγωνιστούμε για κάποια από τα θετικά στοιχεία αυτή τη έκθεση. Ξέρω ότι ο κύριο Σμιτ είναι στην επιτροπή ΕΚΟΝ. Εγώ είμαι αναπληρώτρια εκεί. Αλλά νομίζω πως κάποιες φορές στη σκληρή μας δουλειά σε αυτή την Επιτροπή, όταν πάει στην Επιτροπή, ε, χάνεται και η προστασία του καταναλωτή είναι μια πτυχή που πρέπει να, προστατε... να λαμβάνει την υπόψη πάντα. Πώς θα το κάνει αυτό η συγγετής. Μάλιστα. Ναι, όχι, σωστή η παρατήρησή σας. Όντω πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο κύριος Βίλαν θα είναι διαθέσιμος για να προωθήσει το θέμα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Επισήμως τι γίνεται, τον προσκαλούν. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς γίνεται επισήμως. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Πολύ σημαντική αυτή η πρόταση και όπως μας είπε και η Κομισιόν στην πρώτη συνεδρίαση είναι ένα παλιό θέμα, επιτέλους ήρθε η ώρα να ενεργήσουμε. Ήταν όπως εκείνο με την περιαγωγή για τα κινητά ε, πολλοί κόσμος ε, δεν του πολύ άρεσε το να βάλουμε, να βάλουμε οροφές και τα λοιπά, ε, όπως ο κύριος Σμίτ και οι φιλελεύθεροι. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι η αγορά λειτουργεί καλύτερα χάρη σε αυτή την παρέμβαση. Τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον και πώς το παρακολουθήσουμε είναι ένα σημαντικό τμήμα της πρότασης. Θα δώσω στην κυρία Βέιζεμπεκ το λόγο να δούμε τι γνώμη έχει για αυτή την συνδεστική και μετά ο κύριο για να κλείσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις πολύ επικοδομητικές συναντήσεις που είχαμε εδώ. Εμείς ε, είμαστε σύμφωνοι συνολικά με τις περισσότερες τροπολογίες ε, να κάνω κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί τη λύση για κάποια από τα σχόλια που εκφράσατε και ιδίως ό,τι αφορά τις αναμενόμενες δυσκολίες, ό,τι αφορά τη διασυνορια... τις διασυνορικές αποκτήσεις. Είναι μια δυνατή λύση. Εμείς από πλευράς Κομισιόν ήμασταν πάντα της άποψης ότι αν η συναλλαγή γίνει άπαξ δεν θα πρέπει να είναι ε, χρονοβόρα. μετά από δύο μήνες μπορεί να είναι ε, δυνατή αυτή η διασυνορική απόκτηση, άρα ένας χρόνος είναι μεγάλο διάστημα. Και σε άλλες επιτροπές που συζητήσαν το θέμα αυτό, ε, η απόφαση ήταν να είναι πιο σύντομη η προθεσμία, άρα αυτό μπορεί να είναι μια λύση. Σε ό,τι αφορά ένα θέμα που εξακολουθεί να εκκρεμεί για τις μικροπληρωμές δηλαδή, μπορώ να καταλάβω ε, το επιχείρημα του κυρίου Μπίλαν ε, και τον ορισμό ε, των μικροπληρωμών, πώς ορίζεται η μικροπληρωμές, ίσως θα μπορούσε να κατατεθεί στην Επιτροπή Έκων μια τροπολογία που να λέει ότι υπάρχει ένα σταθερό ποσό και ένα άλλο που είναι ποσοστό, κλιμακώνεται δηλαδή, είναι κειμενόμενο το υπόλοιπο ποσό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ελάχιστο ποσό, ένα μίνιμουμ ποσό, αυτό που προτείνουμε αρχικά ε, βλέπετε ότι δεν είναι πολύ χαμηλό, είναι το ισοδύναμο μίας πληρωμής ε, που ισοδυναμεί με την πληρωμή 35 ευρώ. Δηλαδή, διατραπεζική προμήθεια είναι αντίστοιχη με αυτό που θα πλήρωνε κάποιος ε, για μια πληρωμή 35 ευρώ. Μπορεί να μην είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις τράπεζες γιατί πολλοί εμποροί ε, θα επιμένουν να πληρώνονται τα μικρά ποσά μετρητά. Και αυτό ίσως οδηγήσει σε προβλήματα με τις τράπεζες, ε, μεγάλε, μεγάλους για τις τράπεζες. Γι' αυτό το ελάχιστο ποσό έχω ακούσει και άλλα επιχείρηματα, ότι παραδείγματος χάρη αν υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό πρέπει να υπάρξει και ένα μέγιστο ποσό που δεν είναι και ε, άκυρος επιχείρημα. Αν κάποιος ε, πληρώνει πάνω από 1000 ευρώ, παραδείγματο χάρη, για μια πληρώνη με κάρτα, μπορεί να υπάρχει πράγματι και ένας, αν θέλετε, ένα διακόπτη ε, όταν ε, το ποσό αυτό είναι κάτω ή πάνω από ένα όριο. Θα το αφήσω πάντως στη δική σας σοφία. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σμιτ, στην ΓΑΜΑ ανταγωνισμό συμφωνούμε, καταλαβαίνουμε, ίσως ε, και εδώ βλέπουμε ότι δεν θέλουν ε, ρύθμιση των τιμών, αλλά μετά από 20 χρόνια η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ανταγωνισμός ε, θεώρησε ότι πρέπει να περάσει η ρύθμιση των τιμών ε, πλέον, διότι καταλάβουμε ότι αν το αφήσουμε στη βιομηχανία ε, δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ελήφθησαν αποφάσεις και υπήρξαν και αποφάσεις για θέματα ανταγωνισμού στο μεταξύ, αλλά καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να προβούμε πλέον σε ρυθμίσεις τιμών να σας πω ότι μετά από κάποια χρόνια θα υπάρξει επανεξέταση, δεν ξέρω αν αυτό σας ανακουφίζει. Είναι φιλόδοξη η δική σας πρόταση, θα δούμε πώς θα προχωρήσει, αλλά είναι καλό, είναι καλό να δούμε τις εξελίξεις των αγορών. Η ισχύουσα νομοθεσία άλλωστε θα πρέπει να προσαρμοστεί, γιατί θέλουμε να μπουν στην αγορά και νέοι παίκτες, να δώσουμε κίνητρα, οπότε αν πάνε όλα καλά ίσως ε, να μειωθεί και η ανάγκη για ρυθμίση των τιμών αν έχουμε είσοδο νέων παικτών στην αγορά, αποτελεσματική. Good. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, ήσασταν ξεκάθαροι. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια για το έργο της Επιτροπής μας. Κύριε Μπίλαν, θέλετε να συνοψίσετε. Κύριος Μπίλαν. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν ε, το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Τελικά, το μόνο που παραμένει σε κρεμότητα είναι η τροπολογία του κυρίου Ντεγιόγκ. Όπως διευκρίνησε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θα έχει κάποιες επιπτώσεις μια τέτοια τροπολογία και μπορεί να μην είναι πάντα σύμφωνες με τις επιθυμίες μας και τις προσδοκίες μας αυτές οι επιπτώσεις. Ίσως απόψε ή αύριο το πρωί να προσπαθήσουμε με ανταλλαγέ ηλεκτρονικών μηνυμάτων να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να σα πω ότι έλαβα και μια πληροφορία ότι οι σοσιαλδημοκράτες δεν ήθελαν να στηρίξουν αυτή την πρόταση. Έχουμε όμως λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας ε, και απόψε. Ίσως φτάσουμε ως εκθαύματος σε μια μαγική λύση, δεν ξέρω. Από ό,τι είδα πάντως όλες τις τροπολογίες τις στηρίζουν ή τέλο πάντων ε, περισσότερες αν όχι όλες τις πολιτικές ομάδες ε, και γι' αυτό περιμένω και την αυριανή ψηφοφορία με ανυπομονησία. Πρόεδρος, Μάλιστα, αύριο, όπως είπα, θα ψηφίσουμε όπως είπαμε, διαφορετική σειρά. Η κυρία Βερνιό θα πρέπει να φύγει άρα. Θα ψηφίσουμε μετά τις δύο ψηφοφορίες, ε, τα single votes και τους τριμερείς διαλόγους, το δικό σας θέμα, γύρω στις 10, ως το πιο κοντά στις 10 η ώρα δηλαδή. Θα ψηφίσουμε λοιπόν πρώτα τη δική σας έκθεση. Σας περιμένω αύριο η ΕΚΟΝ την επόμενη εβδομάδα, στις 20 Φεβρουαρίου, θα εγκρίνει τη δική της έκθεση. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Μπίλαν θα έλθει σε επαφή με τους συνάδελφους από την Επιτροπή ΕΚΟΝ για να περάσουν ε, οι απόψεις μας. Θα πρέπει να δούμε και τι θέση θα ακολουθήσουμε στην Ολομέλεια. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι οι τροπολογίες δεν μας καλύπτουν ε, απόλυτα, θα δούμε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ σήμερα το απόγευμα. Θα συνεδριάσουμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 9. 9 το πρωί, γιατί θα έχουμε την παρουσίαση μια νέα πρόταση τη Κομισιόν για τι παραβιάσεις των τελωνικών διατάξεων και την επιβολή κυρώσεων και για την αξιολόγηση επιπτώσεων μελέτη αντικτύπου. 9 με 10. Και έχουμε και άλλες προτάσεις, οποίε θα ψηφισουμε ταξιδιτικά ταξιδιωτικά πακέτα, e-call, σημαντικά νομοθετήματα λοιπόν θα ψηφίσουμε αύριο και μετά θα έχουμε και την έκθεση Βιν Χόλτσερ σε δημόσια συνεδρίες. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.